je dois donner la parole à Madame Gardiazabal pour introduire cette série d'auditions. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Muchas gracias. Voy a ser muy, muy breve. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα... Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, θα είμαι πολύ σύντομη. Ακούτε τώρα ε, να ακούσουμε λοιπόν τους προσκεκλημένους μας ε, ποιο είναι το ο ερώτημα αυτό και πώς απαντάτε. Είναι η ερώτηση του τονός εκατομμυρίου. Ποιο είναι το απαραίτητο μέσο που ε, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά, τι προσφέρεται καλύτερα, εγγυήσεις, επιδοτήσεις ή δάνεια. Ε, και ταυτόχρονα θα πρέπει κάπως να κάνουμε μια απογραφή ε, για το πώς χρησιμοποιούνται στο παρόν χρηματοδοτικό πλαίσιο τα διάφορα μέσα και πώς μπορούμε να τα προετοιμάσουμε για το μέλλον. Κάθε φορά που γίνεται λόγος για χρηματοδοτικά μέσα, πρώτα απ' όλα επικρατεί άγνοια, διότι εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι να χρησιμοποιούμε τέτοια χρηματοδοτικά μέσα στην εκτέλεση του προπολογισμού και είναι γεγονό ότι είναι όλο και μεγαλύτερη η χρήση του, δεν είναι κάτι το νέο, αλλά όταν γίνεται λόγο για τον προπολογισμό είναι πολύ πιο εύκολο ή πολύ πιο σύνηθε να συζητούμε για επιχορηγήσει, για επιδοτήσει από το δημόσιο κορβανά, γιατί είναι και δημόσιε οι πολιτικέ. Και τώρα ε, που κατατρέχουμε, ε, καταφεύγουμε μάλλον ε, όλο και περισσότερο σε χρηματοδοτικά μέσα, θα πρέπει να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση αν αυτά δικαιολογούνται, αν είναι σκόπιμο ή αν είναι χρήσιμο. Και πολλές φορές θα πρέπει να έχουμε την απαραίτητη πληροφόρηση για να ξέρουμε ποιο είναι εκείνο το μέσο ή το είδος δημόσιας στήριξης που προσφέρεται για το κάθε έργο. Επίση, αυτή η συζήτηση ε, γίνεται και ε, σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική, γιατί πολλές φορές ε, το έχουμε δει, έχουμε ακούσει ότι πρέπει λέει, να μειωθούν οι επιχορηγήσεις και να δίνονται περισσότερα χρήματα από τα χρηματοδοτικά μέσα, διότι τα χρηματοδοτικά μέσα είναι πιο φτηνός τρόπος χρηματοδότηση δημοσίων έργων. Και επιπλέον μπορούμε να έχουμε και μια σχετική απόδοση και εθαρρύνουμε και προσελκύουμε και την ιδιωτική επένδυση. Μπορεί όλα αυτά να ισχύουν, αλλά υπάρχουν κάποια έργα και κάποιες πολιτικές που δεν προσφέρονται εξ ορισμού, που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται αμυγός από κρατικές ε, ή από άλλες ενισχύσεις, όχι δάνεια ή χρηματοδοτικά μέσα. Αυτή λοιπόν η συζήτηση που γίνεται αυτό το καιρό θα πρέπει να δούμε κάθε φορά ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη χρηματοδότηση, ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός ή κάποιο άλλο. Και μία από τις ιδέες λοιπόν που εμείς ε, υποστηρίξαμε ε, στην ομάδα μας είναι να θέσουμε στον κύριο ε, Χόρχε Νούνιεθ Φερέρ και όλη την ομάδα του ΣΕΠΣ να κάνει τη μελέτη και στη συνέχεια να ακούσουμε ε, προσώπους αναπτυξιακής τράπεζας ή πρόσωπο κράτους μέλους που διαχειρίζεται άμεσα αυτές τις πολιτικές και τα κονδύλια, αλλά να ακούσουμε επίσης και άλλου είδους τράπεζες όπως είναι η η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αυτά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, να δούμε, να ακούσουμε πρώτα τη μελέτη και στη συνέχεια τα σχόλια των υπολείπων προσκεκλημένων ε, και φιλοξενουμένων μας. Ευχαριστώ. By cadré par notre rapporteur. Y a-t-il pas quelquefois la tentation, lorsqu'on n'a pas d'argent dans le budget, d'avoir recours à l'ingénierie financière Μερικές φορές έχουμε την δυνατότητα να παρεμβαίνουμε σε επίπεδο σύνθεσης χρηματοδοτικών μέσων έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τους στόχους τους οποίους έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτος ομιλητής ο κύριος Φερέρ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν θα σας παρουσιάσω μια έκθεση, θα σας παρουσιάσω τη λογική των χρηματοπιστωτικών μέσων. Έχουμε να κάνουμε με την εικόνα που έχουν οι περιφέρειες οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα μεικτά χρηματοδοτικά μέσα και θα προσπαθήσω να εξηγήσω λίγο τι είναι αυτά τα μέσα και γιατί τα χρησιμοποιούμε. Τα μέσα αυτά δεν αντικαθιστούν τις επιδοτήσεις. Το θέμα είναι βέβαια πώς κατανέμονται και αν μπορεί κανείς να μοιράσει καλύτερα από τη μία τα, τις επιδοτήσεις και από την άλλη τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει τα μεν με τα δε. Εκτός και αν έχουν χρησιμοποιηθεί επιδοτήσεις όταν δεν θα έπρεπε. Εγώ είχα προετοιμάσει την παρουσίαση, αλλά έχει κάπου χαθεί, δεν βγαίνει, δεν ξέρω. Οι διαφάνειές μου δεν είναι, α, δεν ξέρω αν ήταν χρήσιμες, πάντως δεν είναι στη διάθεσή μου. Εκτός αν μπορείτε να μου τις ξαναβρείτε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες εικόνες θα έλεγα που θα καταστήσουν τα πράγματα πιο απλά για σας. Καταρχάς ποιος είναι ο ρόλος των μέσων αυτών των χρηματοδοτικών. Ε, ακούγονται πολλά θεωρητικά και πάρα πολλές ιδέες γύρω από αυτό. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως, τι κάνουν τα μέσα αυτά. και πού παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σαν παράδειγμα. Θα σας παρουσιάσω με απλό τρόπο το πώς λειτουργεί το σύστημα έτσι ώστε να δείτε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και να καταλάβετε το πώς δουλεύει το σύστημα. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των μέσων και θα τον παρουσιάσω ελπίζω με ξεκάθαρο τρόπο. Δεν θα σας ε, παρουσιάσω έτσι και τα προγράμματα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγγυήσει για δάνεια, αυξήσεις κεφαλαίου, χρηματοπιστωτική υποστήριξη, κατά κάποιο τρόπο ένα είδος συμμετοχή στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, αλλά θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω την λογική που βρίσκεται πίσω από τα χρηματοδοτικά μέσα και τις λεγόμενες εξάντε αξιολογήσεις, εκ των προτέρων αξιολογήσεις. σε ποιο βαθμό αυτές οι αξιολογήσεις είναι χρήσιμες όταν θέλει να χρησιμοποιήσει κανείς κάποια τέτοια μέσα. Μετά θα προχωρήσω σε ορισμένες συγκεκριμένες κομβικές τα χαρακτήριζα συστάσεις και θα μιλήσω για τους τομείς στους οποίους πολλές φορές ακούω και το Κοινοβούλιο να λέει ότι αυτόν τον τομέα πρέπει να τον καλύψουμε, αυτόν όχι, ε, τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να είναι χρήσιμα σε συγκεκριμένους τομείς και όχι σε άλλους και το εύση και τι θα κάνουμε με το εύση και πού θα πάει το εύση. Δεν είναι πασπαρτού τα μέσα αυτά για το αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αυτό εξαρτάται από τη δομή τους. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος τώρα της, των μέσων αυτών. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός λοιπόν δίνει δυνατότητες για εγγυήσει, για δάνεια όπως επίσης και για αυξηση κεφαλαίους. Χρηματοδοτούμε ε, θα έλεγα προγράμματα τα οποία να είναι σε θέση να, να χρηματοδοτηθούν και από τα πιστοτικά ιδρύματα ή όταν δεν είναι να τα βοηθήσουμε να γίνουν. Παρεμβαίνουμε ακριβώς έτσι ώστε να καταστούν τα προγράμματα αυτά, προγράμματα τα οποία θα αποσβέσουν τις επενδύσεις τους και θα φανούν πραγματικά χρήσιμα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα χρηματοδοτικό κενό ε, για τα συγκεκριμένα αυτά προγράμματα. Θα πρέπει να είναι καλά τα προγράμματα αυτά, να αξιολογηθούν ως καλά. Δεν ε, φτάνει να πει κανείς ότι υπάρχει μεν ζήτηση και επειδή υπάρχει ζήτηση θα τα καλύψουμε. Θα πρέπει να είναι και συμβατά με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Μερικές φορές κάποια προγράμματα τα οποία είναι μακράς διάρκειας έχουν προβλήματα και δημιουργούν αμφιβολίες για τις εγγυήσει τις οποίες μπορεί να λάβουν και δεν αρκεί το να συνδυάσει κανείς πιστοτικά ιδρύματα για να διασφαλίσει την χρηματοδότησή τους όταν υπάρχουν άλλου τύπου αβεβαιότητες. Ε, έτσι και αλλιώς τα πιστοτικά ιδρύματα περιορίζουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης και σε συνδυαστικό επίπεδο σύμφωνα με τη Βασιλεία 3. Τώρα, ε, υπάρχει η αξιολόγηση του κινδύνου, εκεί όπου υπάρχει ε, χαρακτηρισμός υψηλού κινδύνου. Το θέμα δεν είναι να διατρέξουμε οικονομικά τον κίνδυνο, αλλά να μειώσουμε τον κίνδυνο και ιδιαίτερα όταν μιλάμε όχι για πραγματικό κίνδυνο, αλλά για αντιληπτό κίνδυνο. Ε, πολλές φορές ε, δεν έχουν τα μέσα στη διάθεσή τους ε, για να αξιολογήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι τράπεζες ένα πρόγραμμα και γι' αυτό δεν χρηματοδοτούν τα προγράμματα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και το ανθρώπινο δυναμικό του εξειδικευμένου που απαιτείται έτσι ώστε να καλύψει την συγκεκριμένη ανάγκη και αυτή τη στιγμή βάλει τη σφραγίδα της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τότε και οι υπόλοιποι χρηματοδότες ξυπνάνε και παρεμβαίνουν και αυτοί. Ένας άλλος, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας για τα δημόσια αγαθά, ίσως έχει κανείς περιπτώσεις όπου απαιτούνται επενδύσεις ιδιαίτερα από που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον δημόσιο τομέα και αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, τότε τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα μπορούν να παρέμβουν και να καταστήσουν τους συγκεκριμένους τομείς πιο ελκυστικούς. Αυτή είναι λοιπόν χοντρικά η λειτουργία. Είναι απλά πράγματα, δεν χρειάζεται να μπερδευτούμε ακόμα περισσότερο, Αυτή είναι οι βασικοί κανόνες βλέπετε ε, στις κοκκίδες, βλέπετε τα προγράμματα που είναι τα κόκκινα, τα οποία δεν χρηματοδοτούμε γιατί δεν είναι χρήσιμα για την κοινωνία. Βλέπετε όμως κάποια κίτρινα dots, κάποια κίτρινα κυκλάκια, κουκίδες, που ε, μπορεί να είναι οικονομικά συμφέροντα, αλλά δεν είναι υψηλής χρησιμότητας για την κοινωνία. Τα μπλε ε, είναι αυτά τα οποία καλύπτουν τις ε, ανάγκες της αγοράς. Είναι δηλαδή τα προγράμματα που είναι καλά αλλά δεν έχουν για διάφορους λόγους την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Και εδώ το δημόσιο συμφέρον είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη και όχι συνολικά το θέμα της λειτουργίας των αγορών. Είναι σημαντικό βέβαια γιατί μιλάμε για την αδυναμία των αγορών και όταν μιλάμε για αδυναμία των αγορών στην ουσία λειτουργεί σαν αιτία για ένα κενό, για μια μη ύπαρξη ενός τμήματος της αγοράς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κενό. Βλέπω πάρα πολλές αναλύσεις οι οποίες ε, να προσπαθήσουν να αποδείξουν τη χρησιμότητα των χρηματοδοτικών μέσων. Το θέμα δεν είναι η αιτία των κενών αυτών, το θέμα δεν είναι το μέγεθος των κενών αυτών. Το θέμα είναι να μην κάνει κανείς το λάθος και αντί να καλύπτει τις αδυναμίες της αγοράς, καλύπτει τα αποτελέσματα των κακών πολιτικών που οδήγησαν το ρήγμα αυτό, το κενό αυτό στην αγορά. Αν λοιπόν δεν διορθώνεται το πρόβλημα που δημιούργησε το κενό στην αγορά, <coughs> δεν έχει νόημα να υπάρξει χρηματοδότηση. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει και καταχρήσεις σε τμήματα του πιστοτικού τομέα. Το θέμα δεν είναι το πόσα χρηματοδοτικά μέσα έχει στη διάθεσή σου, το θέμα είναι να μην εξυπηρετείς κακές πολιτικές. Λοιπόν, τώρα κάποιες, κάποιοι βασικοί τρόποι για να μπορέσει να συνεχίσει κανείς. Για την έρευνα και τα μεγάλα προγράμματα υπάρχουν εγγυήσεις για δανειοδοτήσεις, υπάρχουν εγγυήσει για αυξήσεις κεφαλαίων και υπάρχει επίσης και παρέμβαση είτε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είτε του Στρατηγικού Ταμείου ΕΦΣΥ μπορεί να είναι και το Connecting Europe Facility ε, είναι θα έλεγα τα κεντρικά μέσα. Υπάρχει επίσης ένα σύστημα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων και εδώ έχετε πάντα εγγυήσει αυτή τη ε, δυνατότητας ε, έβρεσης κεφαλαίων, δανείων και εδώ παίζουν ρόλο προγράμματα όπως το ΕΦΣΥ, το ΚΟΣΜΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι διαχειριστικές αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να εκδώσουν την δική τους ε, έκθεση εφικτότητας. Και αυτό επίσης περνάει μερικές φορές και από τους οικονομικούς ενδιαμέσους ή χρηματοδοτικούς ενδιαμέσους που είναι οι ιδιωτικές τράπεζες. Και υπάρχουν επίσης και τα διαφθορτικά ταμεία όπως τα ταμεία Urban, επίσης ε, ε, και το ESI που δίδουν εγγυήσεις, δίδουν δάνεια, δίνουν δυνατότητες έβρεσης κεφαλαίων. Ε, αυτές είναι οι τρεις ε, βασικές, ε, αν θέλετε, μορφές χρηματοδότησης τις οποίες μπορεί να βρει κανείς στα πλαίσια των μέσων αυτών. Να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν βρίσκει τα χρήματα αυτά κάπου στον ουρανό αλλά δανείζεται ε, εκδίδοντας ε, ομολογίες και οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας εξαρτάται από το πόσο καλά είναι τα προγράμματα. Χρησιμοποιεί τα ομόλογα για να βρει χρήματα και γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία και η αξιολόγηση μιας τέτοιας τράπεζας. Τώρα για την διαμόρφωση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Στην περίοδο 14-20 βλέπετε ότι καλύπτουμε όλους τους θεματολογικούς τομείς, όλους τους στόχους. Οι διαχειριστικές αρχές μπορεί να φτιάξουν τους δικούς τους τομείς. Ε, υπάρχουν υποχρεωτικές αξιολογήσεις, εκ των προτέρων αξιολογήσεις. Ε, διερευνήσαμε 40 από τις 111 αξιολογήσεις που είχαν γίνει μέχρι το 2015 ε, δεν ήταν εύκολο να βρούμε τις αξιολογήσεις αυτές, ε, δεν είναι διαθέσιμες, ε, δεν είναι διαθέσιμες στην ολότητά τους, στο σύνολό τους. Επίσης είναι και μεγάλου μεγέθους, οπότε είναι δύσκολο να τα εξηγήσει κανείς εύκολα και να κατανοήσει το τι έχει γίνει, ελείπουν και τμήματα και είναι και δύσκολο να βρει κανείς και την μελέτη των επιπτώσεων. Έχουμε λοιπόν εμείς καλύψει περίπου το 50% των <clears throat> αξιολογήσεων που έχουν γίνει. Αν η διαχειριστική αρχή στρέφεται σε κεντρικά μέσα χρηματοδότησης, τότε τα χρήματα δίδονται μεν, αλλά δίδονται μέσω ε, ενός ε, ενδιαμέσου. Και σε αυτή την περίπτωση η εκ των προτέρων αξιολόγηση δεν είναι υποχρεωτική. Το θέμα είναι να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κανείς την αξιολόγηση που έχει γίνει σε κεντρικό επίπεδο και να μην χρειάζεται να δημιουργηθούν επικαλύψεις. Όταν βλέπει κανείς τις αξιολογήσεις αυτές βλέπει ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε αποτυχία της αγοράς. Έχουμε πάρα πολλά έγγραφα που περιγράφουν ακριβώς αυτό που ονομάζουμε market failures, ε, ε, αποτυχημένες μορφές λειτουργίας της αγοράς και υπάρχουν ε, και στοιχεία χώρα αναχώρα. Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς εκ νέου ε, μελέτες. Εγώ βρίσκω ότι το κομμάτι αυτό έτσι και αλλιώ είναι <clears throat> θεωρητικό λιγάκι. Τώρα για την προστιθέμενη αξία, κειμενόμενα τα στοιχεία, μόχλευση, ε, καλά πήγαν τα πράγματα. Τα μαθήματα από το παρελθόν δεν είναι πολύ ικανοποιητική η εκμετάλλευσή τους πολλές φορές τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι χαμηλά. Εμείς ας πούμε λέμε, ξεκινάμε λέγοντας ότι θα δώσουμε 200 δάνεια και στο τέλος είμαστε κοντά σε αυτό έχοντας όμως θέσει ένα πολύ χαμηλό στόχο. Πολλές φορές λοιπόν βάζουμε κάποιους κεντρικούς στόχους οι οποίοι όμως είναι συγκυριακοί. Ε, πολλές φορές υπάρχουν ε, ελλείψεις στον τομέα των αξιολογήσεων από πλευράς των, ε, κρατικών αρχών. Υπάρχουν επίσης πολλές φορές ελλείψεις στον τομέα της ενημέρωσης που δεν επιτρέπουν διορθώσεις της λειτουργίας. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι τα συμπεράσματα αυτά των αξιολογήσεων είναι χρήσιμα, αλλά όχι συνολικά. Πολλές φορές ε, είναι υπερβολικές οι απαιτήσει, χρειάζεται κανείς να περιγράψει μια ολόκληρη σειρά νομοθετήσεων με εκατοντάδες σελίδες ε, και πολλές φορές όταν γίνεται αυτό σε περιφερειακό επίπεδο είναι κάτι που γίνεται και κεντρικά και ασχολούμαστε με τα μη σημαντικά. Το θέμα είναι να δούμε ακριβώς αν υπάρχει κενό στην αγορά, αν υπάρχει μια σωστή στρατηγική επένδυσης και να δούμε ποια είναι τα τελικά αναμενόμενα αποτελέσματα. Τώρα για τη στρατηγική μας, ε, η επενδυτική στρατηγική αυτό έχει σημασία. Πάρα πολλοί σύμβουλοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι, δεν είναι οικονομολόγοι, είναι οικονομολόγοι μάλλον και αξιολογητές, αλλά δεν είναι στρατηγικοί αν θέλετε ε, σύμβουλοι, δεν ε, βλέπουν την πολύ μεγάλη εικόνα. Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών τους δεν είναι πάντα ικανοποιητικά. Βέβαια είναι εύκολο να τους κάνουμε κριτική από τη μία αλλά πρέπει να τους διατηρούμε. Το θέμα είναι ότι αν οι διαχειριστικές αρχές θέλουν να έχουν τους δικούς τους αξιολογητές ε, τότε μπορούν να μην τους χρησιμοποιούν. Αλλιώς όμως αν θέλουν κεντρικά στοιχεία σύγκρισης τότε είναι απαραίτητη. Τώρα για τα συμπεράσματα ανάμεσα σε, σε διαμοιρασμό ευθυνών και σε κεντρικό προγραμματισμό. Να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα μέσα δημιουργήθηκαν, σχεδιάστηκαν ένα ή δύο χρόνια πριν έχουμε στη διάθεσή μας το στρατηγικό ταμείο. Έχουμε λοιπόν αρκετές επαναλήψεις, έχουμε αρκετές ανακατανομές τομέων ανάμεσα σε γενικές διευθύνσεις, στόχους περιφέρειες, επικαλύψεις και πάρα πολλές φορές ε, τα μέσα και στις δύο περιπτώσεις ε, κάνουν τα ίδια πράγματα με διαφορετικές υπηρεσίες και πρόσωπα. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, μπορούμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Αυτό γίνεται, αλλά απαιτείται εξορθολογισμός. Πώς θα γίνει ο εξορθολογισμός. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Είναι αλήθεια όμως ότι τα, χρηματοδοτικά, τα μέσα μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα σε ένα επίπεδο κεντρικού προϋπολογισμού. Να μην υπάρχουν περιφερειακά τέτοια ταμεία. Ε, λειτουργούν σαν ασφάλεια. Αν έχει ένα χωριό και ασφαλίσεις όλα τα σπίτια από μία πλημμύρα ε, και έρθει η πλημμύρα και γκρεμιστούν όλα τα σπίτια θα γκρεμιστεί και ασφαλιστική εταιρεία. Πρέπει να υπάρξει μια κατανομή λοιπόν των εγγυήσεων κατά ποσοστό. Όσο μικρότερο το ποσοστό τόσο υψηλότερη η κάλυψη. Και γι' αυτό ακριβώς είναι καλύτερο να έχει κανείς ένα κεντρικό ταμείο, ο οποίος όμως ένα κεντρικό κέντρο αν θέλετε ε, προγραμματισμού και αξιολόγησης, αλλά αυτό να κατανέμεται ε, αναπεριφέρεια και να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο αυτά τα οποία δεν έχει νόημα να γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω ότι η επόμενη περίοδος λοιπόν είναι ακριβώς η προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτών των μέσων ε, σε κάτι το οποίο να είναι ορθολογικό. Ελπίζω να μην μεσολαβήσουν και άλλες κρίσεις οι οποίες να μας αναγκάσουν να δημιουργήσουμε επιπλέον μέσα. Το θέμα είναι επίσης να δούμε ποιοι είναι οι τελικοί στόχοι. Να μην περιοριστούμε στους ενδιάμεσους στόχους. Αν εκπαιδεύουμε συνέχεια κόσμο, σαν παράδειγμα, στο τέλος θα καταντήσουμε να τους εκπαιδεύουμε για πράγματα για τα οποία δεν χρειάζονται πια. Ε, επίσης και για τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις ε, θα πρέπει να μην δημοσιεύονται μόνο σε ένα κεντρικό μέσο, αλλά θα πρέπει τα, ε, οι αξιολογήσεις αυτές να λειτουργούν κάπως ε, μηχανικά θα έλεγα, να έχουν ένα στάνταρτ διατύπωσης έτσι ώστε να είναι ε, ευανάγνωστα και εκμεταλλεύσιμα εύκολα. Τώρα για κίνδυνος και μη κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αν θα πρέπει να διατρέξει υψηλότερου κινδύνου επενδύσεις ή όχι. Το θέμα δεν έχει σημασία αν είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή οι Εθνικές Επενδυτικές Τράπεζες. Το θέμα είναι να προωθήσουμε προγράμματα τα οποία έχουν προστιθέμενη, υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια από αυτά τα προγράμματα μπορεί να έχουν υψηλό κίνδυνο, κάποια μπορεί να έχουν υψηλή μόχλευση, κάποια μπορεί να χρηματοδοτηθούν εφάπαξη ή συστηματικά, κάποια προγράμματα είναι μακρόχρονα και αυτό κοστίζει. Οπότε το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε στο τέλος ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η μόχλευση από μόνη της δεν είναι ε, το βασικό κριτήριο, ούτε καν το αν είναι κάτι υψηλού κινδύνου ή όχι. Το θέμα είναι να καλύψουμε το τομείς ο οποίους υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Είναι δύσκολο βέβαια να υπάρχουν ε, τέτοιου είδους χρηματοδοτικά μέσα σε πράγματι περιοχές υψηλού κινδύνου. Απαιτείται στήριξη και απαιτείται κεντρικός προϋπολογισμός υψηλού επίπεδου. Το θέμα είναι πώς μπορεί να λειτουργήσει κανείς σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δεν μπορεί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές διαφορετικού επίπεδου κινδύνου. Απαιτείται μια ισορροπία ανάμεσα στα διαθέσιμα μέσα και στη μόχλευση. Όσο πιο ψηλός ο κίνδυνος, τόσο χαμηλότερη μόχλευση. Όσο υψηλότερα τα επιτόκια, τόσο υψηλότερες οι εγγυήσεις που απαιτούνται. λοιπόν, όσο πρέπει να διευρύνουμε τα μέσα, τόσο θα πρέπει και να τα ανασχεδιάζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες του τομέα στον οποίο παρεμβαίνουν. Δεν αρκεί να λέμε ότι ένα μέσο θα πρέπει να αναλάβει και άλλους τομείς. Το θέμα είναι να είμαστε βέβαιοι αν μπορεί να προσαρμοστεί το συγκεκριμένο μέσο αυτό για να καλύψει ένα νέο τομέα. Merci. Ευχαριστώ. éclairage. Ευχαριστούμε για αυτή την κατατοπιστική παρουσίαση. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους και πώς να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όταν ο προϋπολογισμός ε, είναι σε ένα άκαμπτο πλαίσιο, ένα κορσέ. Είδαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. Έπρεπε να καλυφθεί ένα έλλειμμα ε, επενδύσεων. Από τον προπολογισμό δεν γινόταν γιατί το ταμείο ήταν μία. Και πήραν λεφτά από το Connect Europe, από τον ορίζοντα 2020 και βάλαν και στον κουμπαρά μια μαγιά για να προσελκύσουν ε, ε, δάνει και να υπάρχουν εγγύησει των δανείων σε περίπτωση κακοτυχίες. Έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα αρχίσει από τώρα η συζήτηση, κυρία Γκορδία Θάμπαλ. Να περάσουμε ε, στο δεύτερο μιλητή μας. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Ντάβιτ Ντέντσαρ Σπέκ. Um, uh, κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, κύριε Συγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ σήμερα να μιλήσω. Λέγομαι David Tenser Σπέκ και είμαι επικεφαλής του τοπικού γραφείου του KFW που είναι ε, Τράπεζα Πρόθεσης Επενδύσεων της Γερμανίας. Θα σας μιλήσω σήμερα εκ μέρους ε, του οργανισμού που εκπροσωπώ. Το πρώτο όμως που θα ήθελα να αναφέρω ε, είναι ότι όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχει κάποιο είδος εθνικό τράπεζα ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματο που προωθεί τι επενδύσει. Μπορεί να υπάρχουν και δύο ή τρία. Στη Γερμανία έχουμε και περιφερειακά τέτοια ιδρύματα. Να έχετε λοιπόν κατά νου ότι υπάρχουν τέτοιες δομές σε σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο πράγματα θέλω να πω καταρχάς. Να σας εξηγήσω την προοπτική μας. Εμείς ε, παρέχουμε χρηματοδοτικά μέσα στη Γερμανία, αλλά και στη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, θέλω να σας εξηγήσω γιατί δραστηριοποιούμαστε και γιατί θεωρούμε στρατηγικά σημαντικό να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους εταίρους μας στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Πρώτα θα σας μιλήσω για τον οργανισμό που εκπροσωπώ. Κατόπιν θα σας πω λίγα λόγια για το πώς βλέπουμε εμείς τα χρηματοδοτικά μέσα, ποιες είναι οι εμπειρίες μας από αυτά και κάποιες συστάσεις πολιτικής για την περαιτέρω συζήτηση. Ιδρυθήκαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως KFW και βασικός σκοπός ε, του οργανισμού μας ε, ήταν η κατανομή του Ταμείου Μάρσαλ. Και η διαφορά της Γερμανία από άλλα κράτη τη Ευρώπη είναι ότι ε, δεν δώσαμε επιχορηγήσεις όπως, τα όπως οι περισσότερες χώρες, αλλά το κάναμε για να επιχορηγήσουμε δάνεια. Και Νομίζω ότι τα μία Μάρσαλ τώρα κλείνουν τα 70 τους χρόνια και συνεχίζουν να αποτελούν μέρος των κεφαλαίων της Γερμανίας ε, και ανέρχονται πια σε 500 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 70 δισεκατομμύρια ε, αντιπροσωπεύουν τη χρηματοδότηση ε, ενός έτους. Σε σχέση λοιπόν με τους εταίρους μας ε, βρισκόμαστε λίγο πολύ στο, στα ίδια επίπεδα. Μπορεί να πετύχει κανείς μακροπρόθεσμα αποτελέσματα με ε, αυτό το, τον μηχανισμό και θα θέλαμε να συστήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, όταν συμβολεύουμε άλλες χώρες ή παρέχουμε τεχνική βοήθεια για την οικοδόμηση ανάλογων δομών. Αυτό που λέμε είναι ότι απαιτείται χρόνος. Δεν φτάσαμε στα 500 δισεκατομμύρια μέσα σε πέντε χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν μακροπρόθεσμα να προβλέψει κανείς για να πετύχει τέτοια θετικά αποτελέσματα. Χρειάζεται χρόνος για να οικοδομήσει κανείς τις απαραίτητες δομές και για να γίνει αυτό σωστά. Ε, ένα προϊόν παρέχουμε μόνο, την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ απλή δομή. Είναι πολύ απλό αυτό, δεν παρέχουμε υπηρεσίε συμψηφισμού ή πληρωμών. Παρέχουμε μόνο μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά μέσα. Όσον αφορά, όσον αφορά το παθητικό μας, ε, χρηματοδοτούμαστε από τις κεφάλαια αγορές και έτσι ε, μας ενδιαφέρει και εμάς να διατηρήσουμε την ε, αξιολόγηση τριπλό αλφα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να δυσκολεύεστε να διαβάσετε τα γράμματα τα ψηλά σε αυτή τη διαφάνεια, πάντως εδώ βλέπετε τους τομείς ε, στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Στα αριστερά έχετε την χώρια προώθηση επιχειρηματικότητα σε 50 δισεκατομμύρια το χρόνο περίπου, από τη μία προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και από την άλλη προς ε, ε, δημοτικές και ιδιωτικέ επιχειρήσεις. Δεξιά έχουμε περίπου 20 δισεκατομμύρια διεθνή χρηματοδότηση και αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Χειριζόμαστε λοιπόν και τα επίσημα αναπτυξιακά δάνεια της Γερμανίας. Τρία πράγματα θέλω να πω για τη διαφάνεια αυτή. Καταρχάς, ε, εάν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσετε τι κάνουμε ακριβώ. Προωθούμε μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, προωθούμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, έχουμε λοιπόν σαφεί στόχου πολιτική, κάτι που δεν θα πρέπει να σα εκπλήσει. Εφόσον ακολουθούμε κατευθυντήρε γραμμέ τη ομοσπονδιακή μα κυβέρνηση. Υπάρχει επίση συνάφεια ανάμεσα σε αυτά που κάνει η Ομοσπονδιακή μα κυβέρνηση και σε αυτά που γίνονται ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε σε μεγάλο βαθμό του στόχου πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη παρατήρηση, είμαστε ενιαία θηρίδα στην Γερμανία. Σε άλλες χώρες μπορεί κανείς, και να σας δώσω για παράδειγμα τη Γαλλία, μπορεί κανείς να έχει άλλον οργανισμό για την ε, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να έχει άλλον οργανισμό για ε, την χρηματοδότηση δημοτικών υποδομών και άλλον οργανισμό για την χρηματοδότηση των ε, αναπτυξιακών ε, πολιτικών. Στη Γερμανία, λοιπόν, ένα οργανισμό θα έχει αναλάβει όλα αυτά. Σε άλλα κράτη-μέλη μπορεί να έχουμε διαφορετικού οργανισμού. Ποιο είναι το μήνυμα για εσά. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, βρίσκει πάντα τον πιο κατάλληλο εταίρο εντός της χώρας, κάτι που ε, διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Εμείς κάνουμε όλα αυτά στη Γερμανία. Συνήθως όμως ε, δεν χειριζόμαστε μέσα μικροχρηματοδότησης. Για κάτι τέτοιο λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσετε άλλον εταίρο. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό, δηλαδή ε, κατά τη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να βρει κανείς ε, τον ε, κατάλληλο εταίρο. Είτε μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε για κάποια, κάποιον διεθνή οργανισμό προώθησης της επιχειρηματικότητας και υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους διάφορους φορείς, έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το ποσοστό χρηματοδότησης ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσοστό εθνικής χρηματοδότησης. Ε, τρία δισεκατομμύρια λαμβάνουμε περίπου για επιχορηγήσεις από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, 70 δισεκατομμύρια δίνουμε ε, σε κεφάλαια και δάνεια και λαμβάνουμε περίπου 3 δις το χρόνο από, την, από τον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό. Κάτι που δείχνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δεν αποτελούν τη λύση για όλα. Έχουμε διάφορες ε, συζητήσεις ε, με ενδιαφερόμενους κύκλους που θεωρούν ότι μπορούμε να ε, αντισταθμίσουμε τις απώλειες από το Brexit δημιουργώντας περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια σε κάποιο βαθμό. Χρειάζεται όμως και ανάλογη στήριξη από τον προπολογισμό σε διάφορους τομείς. Και για ε, τον ε, οργανισμό μας για το KFW, ε, κάτι τέτοιο θα αντιστοιχούσε σε 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. 70 δισεκατομμύρια χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο για να επενδύσουμε επιχειρήσεις και Είτε επωφελούμαστε από υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε γίνεται απευθεία από την Ευρώπη. Είναι ανάλογο το πώ ε, τα υπολογίσει κανεί, αλλά γενικά δραστηριοποιούμαστε σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε όμω να υπάρχουν πλεονεκτήματα από τη συνεργασία με διάφορους ε, ενδιαφερομένους φορείς της Ευρώπης. Και η τελευταία μου παρατήρηση για τη διαφάνεια αυτή είναι ότι στα αριστερά, αν δημιουργήσουμε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αυτό διαφέρει πολύ από το τι θα κάνουμε στα δεξιά, δηλαδή αν χρηματοδοτήσουμε για παράδειγμα ένα εργοστάσιο παραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας στην Αφρική. Όπως είπα πριν, έχουμε διάφορα είδη μέσων στο ευρωπαϊκό πεδίο. Πάντα πρέπει να βρίσκει κανείς την ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των μέσων που χρησιμοποιεί, κάτι που εξαρτάται και από τον αριθμό των τομέων στον οποίο θέλει να δραστηριοποιείται κανείς. Και η χρηματοδότηση δήμων διαφέρει από την χρηματοδότηση προγραμμάτων ανάπτυξης, για παράδειγμα. Now, um, to the point what we consider τι θεωρούμε χρηματοδοτικό μέσο. Στο εσωτερικό επίπεδο είχαμε μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς ε, θεωρείται χρηματοδοτικό μέσο και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο να το εξετάσουμε από την προοπτική του τελικού δικαιούχου. Λέμε λοιπόν ότι πρόκειται για χρηματοδοτικό μέσο όταν ο τελικός δικαιούχος ε, λάβει επιχορήγηση, δάνειο, ε, εγγύηση κλπ. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν μπορεί να λαμβάνεται υπό μορφή επιχορήγησης, το βλέπουμε αυτό στην αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε ε, επενδυτικές επιχορηγήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που συνδυάζεται από τη δική μας πλευρά με δάνειο προώθησης επιχειρηματικότητας. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι δεν παίζει ρόλο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει την εγγύηση. Αυτό πάντα εξαρτάται από το είδος του μέσου, αλλά ε, τελικά σημαντικό είναι ο τελικός δικαιούχος λαμβάνει επιχορήγηση ή λαμβάνει χρηματοδοτικό μέσο. Όσον αφορά το τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω τέτοιων ε, χρηματοδοτικών μέσων, αυτό ε, έχει να κάνει με την ροή των χρημάτων. Ω ε, άνθρωποι που διαμορφώνονται την πολιτική, λοιπόν, όταν αναρωτιόσαστε αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε επιχορηγήσει ή χρηματοδοτικά μέσα, ε, γενικά είναι σοφό τα χρηματοδοτικά μέσα να δίδονται σε τομεί όπου θα υπάρξει η ροή χρημάτων στο μέλλον. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι φοιτητικά δάνεια, διότι στο μέλλον ο φοιτητής αναμένεται να έχει κάποιο εισόδημα. <laughs> Αναμένεται ότι κάποιος ε, που ε, λαμβάνει ανώτατη εκπαίδευση σε κάποια χρόνια θα έχει μεγαλύτερο εισόδημα. Ε, ε, ανάλογο παράδειγμα είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις υποδομές, εδώ ε, ποικίλει η κατάσταση. Για παράδειγμα, αν χρηματοδοτήσει κανείς εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιήσει χρηματοδοτικό μέσο. Χρηματοδοτούμε όμως και προγράμματα στην Αφρική, όπου εξαρτάται, μπορεί να υπάρχει κάποια ε, δομή πληρωμής τελών. Οπότε να δημιουργείται εισόδημα για να αποπληρωθεί το δάνειο. Πολύ συχνά πρόκειται για πολιτικής φύσης απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθείτε. Γνωρίζετε ότι το θέμα του ύδατο ήταν σημαντικό θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν για πολιτικού λόγου δεν θέλετε να πληρώνονται τέλη για το νερό, εάν θεωρείτε ότι είναι ε, δημόσιο αγαθό το οποίο θα πρέπει να διανέμεται δωρεάν, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματοδοτικό μέσο. Από την άλλη, εάν θεωρήσετε ότι θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε δρόμους, ε, θα πληρώνονται τέλη για το δρόμο, για τη γέφυρα ή οτιδήποτε τότε θα υπάρχει η ροή χρημάτων και μπορείτε να χρηματοδοτήσετε ένα τέτοιο έργο με χρηματοδοτικό μέσο. Να σας δώσω κάποια ακόμη παραδείγματα. Χρηματοδοτούμε σχολική εκπαίδευση για ε, σύρους μετανάστες, κάτι που γίνεται με επιχορήγηση, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, αυτό να, γίνει να αποπληρωθεί στο μέλλον. Επίσης, το άλλο που κοιτάμε είναι η βιωσιμότητα. Και δεν μπορούμε να δίνουμε χρηματοδοτικά μέσα σε κάποιον που δεν περιμένουμε να το αποπληρώσει στο μέλλον. Ε, Στις ε, λιγότερο αναπτυγμένε χώρες, για παράδειγμα, λέμε ότι χρειάζεται επιχορήγηση και αυτό είναι κάτι που αναλαμβάνουν άλλοι φορείς. Τέλος, υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους τομείς ε, δραστηριότητάς μας. Για παράδειγμα, συνήθως δεν χρηματοδοτούμε μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, θεωρούμε ότι έχουν αρκετή πρόσβαση στις κεφαλαίες αγορές Επίσης, ε, όσον αφορά ε, την πλευρά της πολιτικής, θα πρέπει να εξετάσει κανείς ε, αν αναμένονται χρηματικές ζωές στο μέλλον. Τέλος, Εμείς δεν έχουμε ιδεολογική άποψη σχετικά με το αν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτικά μέσα. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και τα δύο. Για παράδειγμα, προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι δεν είναι πάντα γνωστό εκ των προτέρων ε, αν τέτοια μέτρα θα αποδώσουν. Υπάρχουν λοιπόν καλοί τρόποι να συνδυάσει κανείς τις επιχορηγήσεις με τα δάνεια. Άλλο παράδειγμα είναι η αναπτυξιακή βοήθεια όπου υπάρχουν ταμεία που, χρηματοδοτούν είτε μέρος ε, του κεφαλαίου, είτε την εκπόνηση μελετών κλπ. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν το τμήμα που προέρχεται από το προϋπολογισμό της Ένωσης ε, έχει τη μορφή εγγύησης ε, ή δανείου. Ε, σημαντικό είναι τι καταλήγει τελικά στον πελάτη. Εδώ βλέπετε τους τομείς όπου δραστηριοποιούμεθα. Αυτό ισχύει για το KFW, αλλά το ίδιο ισχύει για κάποιους από τους εταίρους μας στην Ιταλία, την Ισπανία και άλλους ε, εθνικούς φορείς και περιφερειακούς. Αριστερά βλέπετε τι κάνουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γερμανία, το COSME, το INOFIN και προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί το κάνουμε αυτό. Καταρχάς μπορούμε να προσφέρουμε πιο ελκυστικά προϊόντα. Λαμβάνουμε ε, κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι παρέχουμε ελκυστικά μέσα χρηματοδότησης. Δεύτερον, μπορούμε να συντονίσουμε ε, την ε, εθνική με την ευρωπαϊκή στήριξη. Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, λοιπόν, συνδυάζουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ε, εθνικό και έτσι έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, σε αντίθετη περίπτωση θα είχαμε αφενός την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου την ε, εθνική πλευρά μέσω του KFW. Αλλά νομίζω ότι γενικά είναι σοφό να δημιουργούμε μέσα που συνδυάζουν τις δύο μορφές χρηματοδότησης. Δεξιά βλέπετε τι κάνουμε στο εξωτερικό, Αφρική, Ασία και Νότια Αμερική. Και εδώ μπορούμε να προσφέρουμε πολύ πιο ελκυστικές προϋποθέσεις στους εταίρους μας στις χώρες αυτές. Εδώ όμως ε, υπάρχει και το θέμα του συντονισμού. Εδώ λοιπόν ο γαλλικός και ο ισπανικός φορέας επίσης δραστηριοποιούνται και όλοι λίγο πολύ ε, ασχολούμαστε με τα ίδια προγράμματα. Έτσι, με αυτόν τον μηχανισμό συνδυασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όλοι συζητάμε, για παράδειγμα, το ίδιο έργο, ε, έναν αγωγό αερίου. Για παράδειγμα, έτσι συζητάμε με τους Ιταλούς και Ισπανούς συναδέλφους μας και ως ευρωπαϊκοί φορείς μπορούμε στις αναπτυσσόμενες χώρες να προσφέρουμε συνδυασμένη χρηματοδότηση για ένα έργο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη μέση βλέπετε την χρηματοδότηση που παρέχουμε στις στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε λοιπόν ε, εθνικούς ε, εταίρους, υπάρχει το Ταμείο Broadband, το Fond που επίσης ε, τρέχει. Ε, ε, χρηματοδοτούμε όμως και εξαγωγές και προγράμματα, κάτι που κάνουμε μόνοι μας και είχαμε και το πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση. Σημαντικό εδώ είναι ότι τα διάφορα μέσα απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες και έτσι έχουν τους δικούς τους κανόνες. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί όταν ε, βλέπουμε ενιαίους κανόνες ε, και, ε, που ισχύουν για όλους, διότι οι συνθήκες διαφέρουν. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη απλοποίησης, υπάρχουν όμως και όρια σε αυτό και υπάρχουν λεπτές ισορροπίες που πρέπει να βρεθούν. Δεν θες να το τελειώσω. Όσον αφορά τις εμπειρίες μας και τις συστάσεις μας. Όσον αφορά τον αριθμό των χρηματοδοτικών μέσων που θα πρέπει να δημιουργηθούν. Για κάθε τομέα πολιτικής πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα. Απ' την άλλη, ε, βλέπουμε κάποιο, κάπως επικριτικά όταν υπάρχουν υπερβολικά πολλά. Για παράδειγμα, έχουμε ένα μέσο που απευθύνεται σε συγκεκριμένε μικρομεσαίες επιχειρήσει στον τομέα του πολιτισμού. Καταλαβαίνουμε την πολιτική ελκυστικότητα του θέματο αυτού. Ε, Ω KFW όμω χρηματοδοτούμε τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει γενικότερα. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, ειδικό μέσο για τον τομέα αυτόν. Εάν χωρίσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει σε 4-5 κατηγορίε ε, μπορεί να γίνουν υπερβολικά πολύπλοκα τα θέματα. Ε, ο λόγος είναι σαφής, ε, κάθε γενική διεύθυνση έχει δικό της προϋπολογισμό. Έτσι λοιπόν είναι ελκυστική η ιδέα του να απευθύνεται κανεί στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά δεν έχει πάντα νόημα μια τέτοια κίνηση. Δεύτερον, ευελιξία. Ε, αν θέλετε να συνεργαστείτε με εθνικούς παραγόντες ελκυστικό και από ευρωπαϊκής πλευράς, θα συνειδητοποιήσετε ότι οι συνθήκες στην αγορά ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό εντός της Ευρώπης. Για παράδειγμα, μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Γερμανία μπορεί να χρηματοδοτείται επί 5 ή 10 χρόνια, ενώ σε άλλη χώρα ε, να απαιτείται χρηματοδότηση μόνο για 3 χρόνια. Όποτε λοιπόν έχει κανείς ενιαίους κανόνες ε, για όλη την Ευρώπη, αν έχουμε δηλαδή 8 χρόνια για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ε, περιορίζουμε τις ε, δυνατότητες για λογική χρηματοδότηση. Συνεχίστε λοιπόν να εργάζεστε με τρόπο ευέλικτο, ώστε να έχουμε 5 χρόνια στην Ουγγαρία, 12 χρόνια στην Πολωνία, 15 στη Γερμανία, 11 στη Γαλλία, ανάλογα με το τι απαιτούν οι συνθήκες της αγοράς. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ε, ότι οι ενιαίοι κανόνε μπορεί να είναι καλοί για μεγάλα προγράμματα υποδομών, αλλά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι εθνικές διαφορές είναι μεγάλες και γι' αυτό ε, έχει πιο πολύ νόημα να έχουμε ευέλικτη προσέγγιση. Όσον αφορά το θέμα της μόχλευσης και της προσθετικότητας, αυτά ήδη αναφέρθηκαν και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, όλοι καταλαβαίνουν Ε, ότι πρέπει να υπάρχουν ε, κάποιοι κοινοί κανόνες και πρέπει να ε, σα συγχαρούμε για τη δημιουργία αυτού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η επιθυμία μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα ήταν να ξεφύγουμε πιο πολύ από το θέμα της ποσότητας και να προχωρήσουμε περισσότερο στο θέμα της ποιότητας. Θα μπορούσαμε να εκπονήσουμε έγγραφο όπου να σας εξηγούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, νομίζω ότι αυτό το γνωρίζει το Κοινοβούλιο, αλλά μόχλευση πετυχαίνουμε όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο αλλάζει και την φύση ενός έργου, διότι πρέπει να αποπληρωθεί και έτσι αποφεύγουμε το λεγόμενο αποτέλεσμα free rider. Αλλά πρέπει πάντα να εξετάζουμε και τους ε, ελέγχους και τα σταθμιστικά μέτρα που είναι απαραίτητα, διότι δίνουμε δάνεια, όχι επιχορήγηση. Εάν δεν πληρώσει κανείς, αυτό είναι αθέτηση υποχρεώσεων. Ο δικαιούχος, λοιπόν, Σημαντικό είναι να λαμβάνει δάνειο ε, με ευνοϊκές προϋποθέσεις, αλλά παραμένει δάνειο. Εάν χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και για τις επιχορηγήσεις, αυτό δεν είναι δίκαιο και δεν θα λειτουργήσει σωστά. Πρέπει λοιπόν να γίνεται η διάκριση ανάμεσα στις επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα. Επίσης, ε, όσον αφορά τους ε, ελέγχους και τα αντισταθμιστικά μέτρα, εδώ δραστηριοποιούνται οι τράπεζες, γι' αυτό θα πρέπει να είναι κάπως πιο ελαφρύ το καθεστώς για τα χρηματοδοτικά μέσα. Ε, νομίζω ότι μπορώ να προχωρήσω πιο κάτω. Βλέπετε εδώ ένα τεχνικό παράδειγμα του είδους των μέσων που χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα όμως να πάω κατευθείαν στην διαφάνεια όπου προσπαθώ να εξηγήσω γιατί συστήνουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, έρχεται σε επαφή με εθνικές τράπεζες ε, προώθησης επιχειρηματικότητας. Ένας από τους λόγους είναι η συμπληρωματικότητα. Αναφέρθηκα και σε αυτό νωρίτερα. Δεν θα πρέπει να θεωρείται επιτυχία το να εξετάζουμε μόνο τις ευρωπαϊκές δυνατότητες στήριξης ή τις εθνικές ή τις περιφερειακές η φιλοδοξία μας θα πρέπει να είναι να εξετάσουμε τις συνδυασμένες δυνατότητες ε, στήριξης για μια μικρομεσαία επιχείρηση σε κάποιον τομέα και να εξετάσουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή εθνικών εταίρων, διότι γνωρίζουν συνήθως καλύτερα τις ε, συνθήκες του πλαισίου, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μικροχρηματοδότηση. Επίσης έχουν πρόσβαση σε εθνικούς πόρους, γνωρίζουν τους τοπικούς παράγοντες και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ε, το, τα δικά μας κεντρικά γραφεία, η δική μας έδρα είναι στη Φραγκφούρτη, αλλά η χρηματοδότηση δίδεται σε στενή συνεργασία με τις περιφερειακές τράπεζες και τις ε, τοπικές τράπεζες προώθησης ε, επενδύσεως. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την γνώση των τοπικών φορέων, των τοπικών τραπεζών που βρίσκονται στην ίδια πόλη με την επιχείρηση αυτοί λοιπόν οι φορεί θα πρέπει να συμμετέχουν για να δημιουργήσουμε καλά χρηματοδοτικά μέσα. Κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Στην KFW αλλά και σε ε, με τους ε, εταίρους μας, συνεργαζόμαστε με ταμιευτήρια, με εμπορικές τράπεζες, Μπορείτε λοιπόν ε, να ε, ε, έρθετε σε επαφή με οποιαδήποτε τράπεζα σε μικρή πόλη μέσω του δικού μας οργανισμού. Και να συνοψίσω τις επιθυμίες μας. Καταρχάς θέλουμε να γίνει καλύτερη χρήση των συνεργειών ανάμεσα στα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα. Δεύτερον, Και αυτό είναι κάτι που ήδη βλέπουμε. Θέλουμε να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στους εθνικούς εταίρους. Ε, έχουμε την αξιολόγηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, των ε, τοπικών ιδρυμάτων. Θέλουμε μείωση της γραφειοκρατίας. Και να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος θέλει δάνειο 100.000 ε, ε, ευρώ για να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να ιδρύσει μια επιχείρηση στη Γερμανία. Μπορεί να λάβει ένα πολύ ελκυστικό προϊόν που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Εθνική Κυβέρνηση και που να μπορεί να πάρει από οποιαδήποτε μικρή τράπεζα. Υπάρχει όμως εδώ ένα μειονέκτημα. Επειδή συμμετέχουν τεσσάρων ειδών φορείς, ε, η KFW, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ε, το Ευρωπαϊκό επίπεδο και το Εθνικό επίπεδο, έχουμε τέσσερι τέσσερις σειρές κανόνων. Πρέπει λοιπόν να υπογράψει κανείς, ε, αλλά το ελεγκτικό συνέδριο, το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο, το KFW και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων πρέπει να λαμβάνει τι σχετικές πληροφορίε ε, που αναρωτιέται κανείς ότι ωραία η χρηματοδότηση είναι μόνο ένα από τα προβλήματα της, νέα ε, νέας μου επιχείρησης. Αξίζει λοιπόν τον κόπο. Χρήσιμο λοιπόν θα είναι να κοιτάξετε όχι μόνο τους κανόνες που επιβάλλετε εσείς, αλλά ε, όλη τη σειρά κανόνων με την οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται ο τελικός δικαιούχος. Εάν καταφέρουμε σε εθνικό επίπεδο να παραλείψουμε, να χαλαρώσουμε κάποιους από τους κανόνες ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ίδιο θα είναι χρήσιμο, διότι πρέπει να εξετάσουμε τον πλήρη κατάλογο των απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρεί ο δικαιούχος. Ε, κατόπιν, ευελιξία και σε αυτό ήδη αναφέρθηκα, οι συνθήκες ε, της αγοράς διαφέρουν από χώρα σε χώρα Χρήσιμο είναι λοιπόν τα ευρωπαϊκά μέσα να έχουν κάποια ευελιξία ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στο εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο. Και τέλος, ε, προβλεψιμότητα. Συνήθως ε, η ευρωπαϊκή συνεργασία στοιχίζει, για παράδειγμα, ε, για τα φοιτητικά δάνεια. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι στο πλαίσιο του Εράσμους. Είχαμε επί δύο χρόνια συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται να επενδύσει κανείς πολύ χρόνο για να δημιουργήσει ένα τέτοιο μέσο. Και στο πλαίσιο του COSME ή του InnoFin, όπου είχαμε ε, τεράστιες επιτυχίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, λέμε ότι θα είναι κρίμα εάν δεν διατίθενται αυτοί οι πόροι μετά το 2020, διότι από τη μία η τραπεζική μας αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν σε τέτοια προγράμματα και μας ενδιαφέρει να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα προγράμματα, εάν αλλάζουν οι κανόνες, εάν υπάρχουν προβλήματα με τον προϋπολογισμό. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα για όλους ε, τους ε, διαμεσολαβητές. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις συστάσεις σας και την έκκληση που απευθύνετε. Ε, για την ευελιξία και τη μεγαλύτερη απλούστευση. Εμείς βουλευτές είμαστε και αφού αυτά τα μηνύματα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ανατόλιο Αλόνσο Πάρδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω, την Επιτροπή σας δηλαδή που μας καλέσατε και είναι ικανοποίηση, ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε την πείρα μας και το όραμά μας από πλευράς μιας διαχειριστικής αρχής. Εμείς ίσως είμαστε πιο κοντά στην ε, πράξη. Ε, θα ε, σας μιλήσω για θέματα πιο χειροπιαστά και πιο πρακτικά. Ελπίζω να σας βοηθήσουν τα σχόλια και οι συστάσεις και οι δικές μας. Είναι πιο πεζά ίσως αυτά που θα σας πω. Σε πέντε τμήματα χωρίζεται η παρουσίασή μου. Μια σύγκριση πρώτα της παραδοσιακής μεθόδου χρηματοδότησης διαφόρων δράσεων από τα διευθυντικά ταμεία που βασικά πρόκειται εκεί για επιδοτήσεις και μετά τα χρηματοδοτικά μέσα. Νομίζω στη συνέχεια θα αναφερθεί η επόμενη ομιλήτρια σε αυτό το θέμα. Επίσης θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τα χρηματοδοτικά μέσα στα ε, επιχειρησιακά προγράμματα της Ισπανίας στην προηγούμενη και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε την άποψή μας για τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις δυσκολίες ε, για τη δρομολόγηση και την εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων, ιδιαίτερα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και μετά θα αναφερθώ λίγο σε κάποιες από τις καινοτομίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός Omnibus, που αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα. Και τέλος, όπως και οι συνάδελφοι, θα σας απευθύνουμε μερικές συστάσεις κι εμείς. Λοιπόν, συνήθως οι δράσεις ε, που χρηματοδοτούνται από τα χρηματοδοτικά ταμεία ε, επιδοτούνται. Δηλαδή δεν επιστρέφεται, δεν είναι δάνειο, είναι επιχορήγηση. Έχουμε δημόσιες ε, επιχειρήσεις που επενδύουν ή που έχουν προγράμματα επιδοτήσεων και βοήθειας και αυτή τη στιγμή εκτελεστεί η δαπάνη που έχει επιλεγεί μας στέλνουν ε, το τιμολόγιο για να αποζημιωθούν. Εμείς τα ελέγχουμε αυτά, τα στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έρχεται η αντίστοιχη βοήθεια. Έτσι είναι η κλασική μορφή χρηματοδότησης μέσω των διορθωτικών ταμείων και πρόκειται εκεί για επιδοτήσεις. Βεβαίως μεταξύ αυτών υπάρχει και επιδότηση ε, επιτοκίου ή τα προτιμασιακά δάνεια, δάνεια δηλαδή με, ευνοϊκό επιτόκιο. Και αυτό επίσης μπορεί να είναι επιλέξιμη δαπάνη. Δηλαδή ένα ευνοϊκό επιτόκιο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς. Και αυτό είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης. Ε, δεν είναι χρηματοδοτικό μέσο, ε, είναι δάνειο και όχι επιχορήγηση, αλλά παρόλα αυτά ε, αντιστοιχεί. Λοιπόν, η άλλη επιλογή είναι το χρηματοδοτικό μέσο. Η διαχειριστική αρχή λοιπόν τι ε, πιστοποιεί. Εμείς πιστοποιούμε τα έσοδα ότι καταβάλει κάποιο ένα ποσό που δίνει εγγυήσει, ε, σε ένα οργανισμό μάλλον που δίνει ε, ε, εγγυήσεις, δάνεια ή συμμετοχικά δάνεια ή διάφορα άλλα μέσα τα οποία έχω ξεχάσει. Πάντως, αυτό είναι η δαπάνη επιλέξιμη από μόνη της. Η συμμετοχή και αυτό πιστοποιείται στη διαχειριστική αρχή. και αυτό στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούμε ε, μια ε, προκαταβολή ή ενδιάμεση πληρωμή. Βεβαίως από εκεί και πέρα το χρηματοδοτικό μέσο το οποίο διαχειρίζεται ένας εκτελεστικός ε, οργανισμός στέλνει τη χρηματοδότηση στο δικαιούχο, ένα από τα τέσσερα αυτά προϊόντα. Και μάλιστα ο κανονισμός κάνει λόγο για τελικό αποδέκτη, όχι δικαιούχο. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα ή έμεσα, μέσω από κάποιο οικονομικό διαμεσολαβητή μεσάζοντας. Η διαχειριστική αρχή λοιπόν που λαμβάνει τη βοήθεια οφείλει να απορροφήσει πλήρως το ποσό και αν υπάρχει ένα ποσό που δεν έχει δαπανηθεί οφείλει να επιστραφεί. Είναι αρκετά διαφορετικός τρόπος διαχείρισης από τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης των επιδοτήσεων. Λοιπόν, τα χρηματοδοτικά μέσα εισήχθησαν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο παρελθόν τα χρησιμοποιούσαμε μένα, αλλά δεν ε, τα ανέφεραν ρητά οι κανονισμοί. Από την προηγούμενη λοιπόν προγραμματική περίοδο που έληξε το 2013, και που στις 31 Μαρτίου ε, στείλαμε όλα τα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε δύο άρθρα του κανονισμού που αναφέρονται ειδικά σε τέτοιου είδους χρηματοδοτικά μέσα. Και στον εκτελεστικό επίσης ε, κανονισμό άλλα δύο άρθρα αναφέρονται σε χρηματοδοτικά μέσα. Στην προηγούμενη περίοδο ε, γινόταν λόγος για ε, χρηματοοικονομική μηχανική. Εγώ και εγώ που είμαι μηχανικός με τρομάζει να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο ε, χρηματοοικονομική μηχανική, να το συνδέω με τα χρηματοοικονομικά. Εν περιπτώσει, αυτά έλεγε ο κανονισμός. Ε, ε, είχε αρκετές ατέλειες και αδυναμίες στην αρχή και ξεκίνησαν δύο πρωτοβουλίες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον Τζέρεμι και τον Τζέσικα. Ε, Το Τζέρεμι ήταν για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η Τζέσικα ε, για την αστική ανάπτυξη και την ενεργειακή απόδοση. Και τέλος, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη. Ε, ποια είναι αυτή να ενισχυθεί η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, δηλαδή να διευκολυνθούν κάπως, ή ε, τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία, δεν ξέρω αν πάντα αυτό γίνεται, ε, κάποια διευκόλυνση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Παράδειγμα, ορίζονται κάποια ε, χρηματοδοτικά μέσα που ε, είναι έτοιμα και μπορεί κάποιος να τρέξει σε αυτά που δεν έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Από την άλλη, ε, υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά μέσα που απευθύνονται σε όλα τα κρατη και τα διαχειρίζεται άμεσα η έμεσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ε, σημαντική καινοτομία. Τώρα δεν βλέπετε τίποτα στη διαφάνεια αυτή, αλλά Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΦΕΝΤΕΡ και τα διαφορετικά ταμεία προτιμούν τι επιδοτήσεις, το κλασικό παραδοσιακό ε, χρηματοδοτικό ε, σχήμα. Το 85% στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο της κοινοτικής βοήθειας ήταν ακριβώς με τη μορφή των επιδοτήσεων. Και μόλις το 15% ήταν δάνεια, ήταν επιστρεφόμενες ε, βοήθειες. Και επειδή ήταν καινούρια αυτή η κατάσταση, ασυνήθιστη, ε, είχαμε και ένα μείγμα χρηματοδότησης, δηλαδή ε, επιδοτήσεις και δάνεια. Με την ατυχία να έχουν τα ίδια και τον ίδιο κωδικό πολλές φορές και οδηγηθήκαμε σε συγχύσεις εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, αν δούμε μόνο το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, το 8% μόλις ε, ήταν δάνεια. Η άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Το 8% μόνο, το υπόλοιπο ήταν επιδοτήσεις. Τώρα, χρηματοδοτικά μέσα στην πράξη. Δεν έχω τη φιλοδοξία να το διαβάσετε αυτό στη διαφάνεια, αλλά υπάρχει και σε έγγραφο και μπορείτε να το εξετάσετε και να το μελετήσετε με την ησυχία σας. Τι βλέπουμε εδώ. Στην περίοδο 2007-2013 διαχειριστήκαμε 14 χρηματοδοτικά μέσα, 12 τύπου Τζέρεμι, αν και από τα 12 αυτά μόνο το ένα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τα άλλα ήταν σε εθνικό επίπεδο, αλλά με την ίδια έτσι, λογική φιλοσοφία, γι' αυτό λέμε τύπου Τζέρεμι ότι ήταν τα έργα αυτά, και συνολικό ποσό είχαμε 230 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων απορροφήθηκαν τα δύο τρίτα. Επίσης είχαμε άλλα δύο μέσα, αυτή τη φορά ήταν τύπου Τζέσικα, όχι Τζέρεμι, γιατί ήταν ε, στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 220 εκατομμύρια ευρώ, 75% απορρόφηση. Μεταξύ λοιπόν των 14 χρηματοδοτικών μέσων συνολικά ήταν 1,5 δις περίπου και απορροφήθηκαν κατά 70% από το ΕΤΠΑ, το ΦΕΝΤΕΡ, τι δώσα μέσα, χρηματοδοτικά μέσα, το, τα μισά από το 8% που σας ανέφερα προηγουμένως. Ένα 4% λοιπόν ήταν επιδότηση επιτοκίου ή δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο ή ε, προνομιακή ε, δανειοδότηση. Τώρα, στην τρέχουσα ε, περίοδο, τι έχουμε κάνει. Το ΕΣΠΑ 800 εκατομμύρια ευρώ από μόνο του είναι χρηματοδοτικό μέσο το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε λοιπόν κεντρική διαχείριση και συνολική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και οι βασικοί χρήστες είμαστε εμεί. Δηλαδή η Ισπανική Διαχειριστική Αρχή ήταν η πρώτη που έκανε χρήση αυτού και αφορά ιδιαίτερα εδώ το άρθρο 39 του κανονισμού κοινών διατάξεων και ουσιαστικά πρόκειται για ταμείο εγγυήσεων. Στη δική μας περίπτωση χρησιμοποιήσαμε ε, τη δυνατότητα εγγυήσεων για νέα δάνεια χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τη διτλοποίηση που και αυτή προβλεπόταν από τον κανονισμό, αλλά ε, ε, εννέα τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έλαβαν μέρος. Και το χρηματοδοτικό αυτό μέσο όταν δρομολογήθηκε γνώρισε μια μεγάλη δυσκολία χρηματοδότησης ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. γιατί σκοπός είναι να χρηματοδοτούνται με ένα γρήγορο ρυθμό και να απορροφάται πλήρως το μέσο μέχρι το 2019, δηλαδή αρκετά ε, νωρίτερα από την περίοδο επιλεξικότητας που κλείνει ε, το Νοέμβριο του 2023. Η ανταπόκριση ήταν πολύ καλή. Ε, τα μπλοκ των εγγυήσεων τώρα έχουν κατανεμηθεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, κατά το 96% και καλύπτεται στη τάξη μεγέθους 4 προς 1 ε, το σύνολο της επικράτειας, εθνικό επίπεδο δηλαδή. Στην Ισπανία αυτή η συμφωνία χρηματοδότησης λόγω της διοικητικής δομής της χώρας και μηχανής χρειάστηκε να προχωρήσει σε κάποιες δεσμεύσεις για κάθε μία από τις 19 αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας. Αυτό το 4 προς 1 δηλαδή ισχύει ε, για όλες τις αυτόνομες περιφέρειες που δεν έχει γίνει πραγματικότητα, έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Ως αποτέλεσμα λοιπόν του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα διευρυνθεί και αυτό το χρηματοδοτικό μέσο και θα έχει πάνω από 117 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Με τις συμβάσεις που έχουν γίνει και τις συμφωνίες με τις τράπεζες, φτάνουμε στα 5,5 δις ε, δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αρκετά ψηλότερο το ποσό σε σχέση με τα νησίοντα στην προηγούμενη περίοδο. Επίσης, δρομολογούμε άλλα χρηματοδοτικά μέσα αυτό τον καιρό έτσι πιο παραδοσιακού χαρακτήρα. Είμαστε στη φάση της ε, εκ των προτέρων αξιολόγησης που είναι και υποχρεωτική, στην οποία αναφέρθηκε ο Και αυτή τη στιγμή προβλέπουμε ε, να ε, ξεκινήσουμε άλλα 17 χρηματοδοτικά μέσα σε περιφερειακό επίπεδο και ένα σε εθνικό επίπεδο. Συνολικά με συντηρητικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς, γιατί δεν έχουμε το τελικό ποστό για τις μικρομεσαίες, θα είμαστε ακόμα σε 1,5 δις. Δηλαδή, σε σχέση με το ΦΕΝΤΕΡ για την Ισπανία διπλασιάζουμε τη χρηματοδότηση ε, συγκρινόμενη με την προηγούμενη πραγματική περίοδο. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πιο περιορισμένους ε, πόρους. Συνεχίζουμε τώρα. Για να δούμε ποια είναι η δική μας αντίληψη για αυτά τα πράγματα, τα υπέρ και τα κατά των χρηματοδοτικών μέσων. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να αναχρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί. Το είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως. Και επίσης είναι και ο πιο κατάλληλος τρόπος να έχουμε δημόσια παρουσία ε, σε περίπτωση κεφαλαίων κινδύνου, συμμετοχικών δανείων ή εγγύησεων. Δεν μπορώ να φανταστώ διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης τέτοιων ε, μορφών. Επίσης, είναι μια εναλλακτική μορφή ε, χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων με βοήθειες υπό τη μορφή δανείου. Δηλαδή, αν έχει αρκετά κεφάλαια κίνησης, ένας ε, οργανισμός μπορεί να δίνει τέτοια δάνεια και να πιστοποιείται αυτό, να το διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, ανταμείβεται, να έχει την απόδοση. Αλλά δεν έχει πάντα αυτή τη ρευστότητα ένας ε, χρηματοπιστωτικός οργανισμός, μια τράπεζα για να δίνει τα συγκεκριμένα δάνεια. Είναι καλή λύση λοιπόν αυτό, καλή δυνατότητα ε, χρησιμοποίησης αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Ε, τέλος, σε πολλές περιπτώσεις, όπως τώρα, το συνολικό ποσό αυξάνεται δεδομένων και των επιδοκίων. Μετά είναι ένας τρόπος γρήγορης εκτέλεσης ε, και απορρόφησης των κοινοτικών πόρων αντί να πιστοποιεί και να εγκρίνεις πρόγραμμα-πρόγραμμα, έργο-έργο, μπορείς να έχεις ένα συνολικό φάκελο, να χρηματοδοτηθεί το έργο και να προχωρήσει πιο γρήγορα. Και αυτό πλέον έκτημα είναι. Το κόστος επίσης τη διαχείριση, το λειτουργικό και το ποσοστό, είναι ένα ε, τμήμα του ε, χρηματοδοτικού μέσου. Δηλαδή, δεν καταναλώνονται πόροι για τεχνική βοήθεια. Δεν χρειάζεται να εγγράψει στον προπολογισμό του έργου επιπλέον τεχνική βοήθεια. Αυτό είναι σημαντικό και ενδιαφέρον ως πλεονέκτημα. Και τελευταίο, σημαντικό, η δυνατότητα να κινητοποιείται ε, ιδιωτικό κεφάλαιο. Και επιπλέον εποφελούμαστε ε, από την ε, εμπειρία του ιδιωτικού τομέα και την διασύνδεσή του με τις τράπεζες. Άλλα πλέον εκτήματα για το 14-20, η δυνατότητα να έχουμε ε, κεντρική διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων. Έχουμε 100% συγχρηματοδότηση, δηλαδή αυτό που σας είπα προηγουμένως το χρηματοδοτικό μέσο για την πρωτοβουλία για τις ε, μικρομεσαίες είναι μηδενική συμμετοχή του κράτου. Αρκεί να πει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποιοι είναι οι πόροι που χρειάζονται, έτσι ώστε η διαχειριστική αρχή να διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζομαι χι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έρχονται αμέσω χωρί να υπάρχει εθνική συγχρηματοδότηση ή αντιστάθμισμα. Θεωρητικά τώρα πάντα όλα αυτά. Επίση υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο το οποίο θα καλύπτει όλες τις πολιτικές μιας προτεραιότητας ε, των διευθυντικών ταμείων. Αυτό έχει ένα πριμ της τάξης των 10% και αυτό ενδιαφέρον στη χρηματοδότηση. Και τέλος, πάντα σε αυτές τις δυνατότητες χρηματοδότηση των ταμείων υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουμε μια ενδιάμεση πληρωμή, μια προκαταβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, προβλέποντας την εθνική συμμετοχή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ε, έρθει η κρατική συμμετοχή από την αρχή, ε, αρκεί και μόνο η δέσμευση ότι θα ακολουθήσει σε ε, ευθετότερο χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχουν εκεί και είναι σημαντικό. Να, υπάρχει δυνατότητα να χαρακτηρίζονται εκτελεστική διαχειριστική αρχή χωρίς να προκηρυχθεί κάποιος διαγωνισμός κτλ. Σας είπα για τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι προκαθορισμένα για όλα τα κράτη-μέλη, είναι δύσκολο όταν σε μια περιφέρεια, σε ένα κράτος αρχίζει να λειτουργεί ένα χρηματοδοτικό μέσο, να ανταποκρίνει σε 100% των off-the-shelf έτοιμων δηλαδή προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων. Τελευταίο άλλο πλεονέκτημα είναι ακριβώς ότι η στοχή της θεματικής συγκέντρωσης της περίοδου 14-20. Ε, έρευνα και ανάπτυξη, στήριξη μικρομεσαίων, ε, τεχνολογία της πληροφορίας ε, και οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ας πούμε για αυτή την τελευταία οικονομία χωρίς διοξιδίου του άνθρακα ξέρουμε ότι για την προσέλκυση επενδύσεων ε, για την ενεργειακή απόδοση ε, προβλέπεται απόδοση. Δηλαδή γίνεται οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας για να μπορέσεις να αποπληρώσεις το δάνειο. Ακριβώς είναι και βιώσιμο και συμφέρει το μέσο αυτό. Αν έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, θα μας ρωτήσετε γιατί είστε μόνο στο 8-9% γιατί δεν έχετε πάει στο 60% αν είναι τόσο ευνοϊκή η κατάσταση. Γιατί θα έρθω τώρα στις δυσκολίες και τα μειονεκτήματα. Βεβαίως, δεν μπορούν όλα τα χρηματοδοτικά μέσα να χρηματοδοτήσουν ε, κάθε ε, δημόσιο έργο. Λοιπόν, έχω εδώ όλα τα αρνητικά τώρα. Είναι περίπλοκο το σύστημα, χρόνο η εκ των προτέρων ε, αξιολόγηση, σύμφωνα με τους οδηγούς και τα λυσάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ εξαντλητική και βαριά διαδικασία όσο και μακροχρόνια και οι διαχειριστικές αρχές, ακριβώς για να μην βρούμε τον πελά μας, είμαστε πάρα πολύ σχολαστικοί στον έλεγχο. Προτιμούμε ε, να τα έχουμε ελέγξει όλα, μην τυχόν και γίνει κανένα λάθος. Βεβαίως ε, οι συμφωνίες χρηματοδότησης που είναι το βασικό εργαλείο που διέπει κάθε χρηματοδοτικό μέσο και θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία με τον εκτελεστικό οργανισμό είναι πάλι πολύ βαριά, αρκετά βαριά διαδικασία. Ειδικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πολύ βαριά γιατί ε, στις διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πάρα πολύ επίμονη, πάρα πολύ σχολαστική. Πάνω από ένα χρόνο χρειάζονται διάφορες συμφωνίες για να υπογράψουμε. Δεν είναι μόνο απλή συμφωνία χρηματοδότησης. Υπάρχουν διάφορες συμφωνίες ε, για την χορήγηση δανείου. Όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία δεν είμαστε εμεί συνηθισμένοι. Και μας παραξένεψε και λίγο. Ήταν αρκετά βαριά και πολύ γραφειοκρατική διαδικασία. Επίσης, οι διαχειριστές δεν έχουν την εμπειρία διαχείριση τέτοιων χρηματοδοτικών μέσων. Εμείς δίναμε χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις για μεγάλα έργα υποδομών ή για καθεστώτα βοήθειας. Στο ΦΕΝΤΕΡ, ας πούμε, δεν είχαμε συνηθίσει τέτοια χρηματοδοτικά μέσα και είχαμε κάποια αρχική, πώς να το πω, ένα δισταγμό, μια φοβία. Κάτι άλλο που δεν είναι ίσονος σημασίας, είναι περίπλοκος ο κανονισμός. Υπάρχει ε, μια καυκική διάσταση, υπερβολική ε, μέρημνα ε, για ρύθμιση. Ήταν λίγα τα άρθρα στην αρχή, ενώ τώρα και μόνο ο τίτλος 4 έχει 10 άρθρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα διαβάσει κανείς και να τα έχει υπόψη του κατεξουσιοδότης κανονισμός ε, και τέσσερις εφαρμοστικοί κανονισμοί και 14 οδηγίες και παραπάνω. Μπορεί να έχω ξεχάσει και καμία ε, και προσανατολισμοί για το πώς θα διαχειριστούμε αυτά, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που είναι και μια παράλληλη ε, νομοθεσία η ρύθμιση, κανόνες. Είναι παρακανόνες, δεν είναι ακριβώς κανόνες, αλλά πολλές φορές έχουν μεγαλύτερη ισχύ και, πιο αυστηρά αποτελέσματα από τον ήταν ένας κανονισμός, ε, κανονικός συνομοθεσία. Και υπάρχουν και πολλοί περιορισμοί κανονιστικοί που δυσκολευόμαστε να τους καταλάβουμε. Υπάρχει μια δυσκολία να συνδυάσουμε τις ε, ε, ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα. Πολύ πρόσφατα είχαμε μια αμφιβολία για το τι εφαρμόζεται, τι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και να συνδυάσουμε. Και ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται συνδυασμός, αλλά στις δύο επόμενες σελίδες ε, καταλήγει ότι αποκλείεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζει. Ενώ θεωρητικά σου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνδυάσεις και επιδοτήσει με χρηματοδοτικά μέσα. Άρα, πού οδηγούμαστε. Έχουμε μια νομική αβεβαιότητα είναι πολλές φορές ήξεις αφήξεις, χρησμοί αυτά που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας πούμε για το κυκλικό κεφάλαιο, για το... Ε, ε, ε επαναχρησιμοποίηση ε, πόρων κλπ. Ε, πραγματικά πολλές φορές ψοκινδυνεύουμε άλλα στοιχεία που έχουν σημασία. Τώρα επαναλαμβάνομαι, αλλά τα χρηματοδοτικά μέσα νομίζω υπερβάλλουν. Είναι περίπλοκα, είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερα προαπαιτούμενα από ένα κλασικό εθνικό χρηματοδοτικό μέσο. Ε, παράδειγμα. Η ενημέρωση, πληροφόρηση είναι εξαντλητική, είναι σχολαστική, είναι πολύ λεπτομερής για τους ελέγχους. Ε, στις επιδοτήσεις ελέγχουμε τη δαπάνη, τη δημόσια δαπάνη. Βλέπουμε αν έχουν γίνει οι επενδύσεις με τη συγκεκριμένη συγγραφή υποχρεώσεων, ότι το έργο έχει αποτέλεσμα. Αλλά εδώ πρόκειται για δάνειο και εκείνο που δίνει το δάνειο θέλει να το ανακτήσει και όλα δείχνουν ότι θα το ανακτήσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν έξτρα προαπαιτούμενα ελέγχων και παλήθευση πολλέ φορέ δεν είναι εύκολο να ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουμε. Για το, για το κεφάλαιο κίνηση ή το κεφάλαιο κινδύνου, ποια χρονική στιγμή θα πρέπει αυτό να το ελέγξουμε. Τη στιγμή που χορηγείται το δάνειο, που εγκρίνεται μετά από δύο χρόνια πότε και τι εγκρίνεται, η δαπάνη που έγινε η επένδυση. Ε, όχι, για αφού ήταν κεφάλαιο κίνηση, ποια επένδυση και τι ελέγχουμε. Και αν δεν συμπίπτει αυτό με το επιχειρησιακό σχέδιο που είχε κατατεθεί στην αρχή, σημαίνει ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί. Μα όλος δάνειο έχει ζητήσει. Δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, πώς να το πω, που απορρέει από το γεγονός ότι ε, κάνουμε μια πολιτική που ακολουθούμε στις επιδοτήσεις για κάτι το οποίο είναι δάνειο και αποπληρώνεται. Εμείς πάντα συστήνουμε στους περιφερειακούς οργανισμούς να συμφωνούν και εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό σε εθνικό επίπεδο με ε, την ε, αρχή που κάνει τον οικονομικό έλεγχο. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο αυτό και να έχει και κινδύνους. Συνέπεια άμεση για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Οι τράπεζες το σκέφτονται πάρα πολύ πριν μπουν ε, σε αυτή την ε, τράπο, σε ένα τέτοιο ε, χρηματοδοτικό μέσο. Και αν θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικό κεφάλαιο, όχι μόνο από την απλή διαμεσολάβηση, δηλαδή να βάλουν και κεφάλαια, μπορεί κάποιος συγκεκριμένος έλεγχος να έχει και συγκεκριμένες συνέπειες, το ξανασκέφτεται το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή που καλείται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Στον οικονομικό συλλογιστικό έλεγχο. Είναι εκ των υστέρων έλεγχος, δεν είναι ο ίδιος εσωτερικός οικονομικός έλεγχος, αλλά είναι ίδιο το αποτέλεσμα, είναι αποθαρρυντικό. και μας οδηγεί στο να ε, επιλέγουμε προγράμματα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε κεντρικό επίπεδο. Γιατί λέμε θα είμαστε περισσότερο καλυμμένοι και ας μην μπλέκουμε τώρα με προγράμματα που θα διαχειριζόμαστε εμείς για να βρούμε στη συνέχεια το μπελά μας. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, αν το χρηματοδοτικό μέσο το, το διαχειρίζεται ένας ενδιάμεσος οργανισμός ή η υπηρεσία που γενικά ε, χειρίζεται τις επιδοτήσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ε, υπάρχει περίπτωση να το διαχειριστεί κάποιο που διαχειρίζεται επιδοτήσει με την ίδια αυστηρότητα και σχολαστικότητα, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Όταν κάποιο θέλει ένα δάνειο, ε, για να προχωρήσει σε μια καινοτόμα δράση χρειάζεται πιο ελαφρές διαδικασίε. Έχω εδώ ένα κατάλογο των μέτρων και των κανόνων που ισχύουν και τελευταίο που θέλω να σας αναφέρω είναι κάποιες καινοτομίες που έχουμε στη νέα πρόταση Omnibus με τον κανονισμό αυτό. Το πρώτο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα πρέπει να δούμε τις δυνατότητες μα είναι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το σχέδιο Juncker. Να δούμε. Αυτό το, το χρηματοδοτικό μέσο ε, είναι κεντρική διαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι 100%, δηλαδή με μηδενική κρατική χρηματοδότηση. Όπω είναι η πρωτοβουλία για τι μικρομεσαίε ε, που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άλλη σημαντική βελτίωση και ενδιαφέρουσα. Δεν χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα για την πρωτοβουλία ε, για τις μικρομεσαίες, αρκεί να είναι προτεραιότητα ενός προγράμματος. Κάτι άλλο που μας ανησυχεί είναι πώς γίνεται ο οικονομικός έλεγχος όταν διαχειρίζεται τα προγράμματα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό μας ανησυχεί γιατί σύμφωνα με τη νέα πρόταση κανονισμού Omnibus εξαιρείται από τις εξάντε υποχρεώσεις ε, έλεγχο και δεν ελέγχεται από τις εθνικές αρχές. Εκεί δεν σημαίνει ότι έχουμε απαραίτητο αντίρρηση, αλλά ανησυχούμε μήπως αυτό χαθεί, δεν μιλώ για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπάρχουν άλλες τράπεζες ή και τελικοί δικαιούχοι που είναι ε, αυτό αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να χαθεί ο έλεγχος από τα κράτη-μέλη. δεν τα διαχειρίζεται πάντα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτά τα δάνεια, αυτά τα έργα. Εκεί μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνο. Δηλαδή εμεί ελέγχουμε κάποια πράγματα που ελέγχει και κάποιο άλλο, ο οποίο εξαιρείται το ελέγχο. Συστάσει. Απορρέουν οι συστάσεις από αυτά που σας είπα μέχρι τώρα. Θα πρέπει τα χρηματοδοτικά μέσα να ε, έχουν ξεχωριστή διαχείριση από εκείνη των διαρθρωτικών ταμείων. Άρα χρειάζεται άλλο σύστημα. Ένα κανονιστικό ρυθμιστικό σύστημα που να τα ορίζει αυτά με τρόπο πάρα πολύ απλό, ρητό και σύντομο και όχι υπερβολική ρύθμιση. Επίσης, δεν θα πρέπει τα δάνεια και οι επιχορηγήσεις να έχουν την ίδια αντιμετώπιση σε σχέση με τον τελικό αποδέκτη δικαιού. Άλλο επιχορήγηση, άλλο το δάνειο. Δυστυχώς τώρα έχουν ευθυγραμμιστεί αυτά. Και επίσης ορισμός της ε, συναλλαγής. Και είναι, η αρχική οικονομική υποστήριξη αλλά και οι μελλοντικέ μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μέσου. Δηλαδή το σύνολο και το υποσύνολο είναι ε, το operation αυτό, η δράση. Δηλαδή κάθε δάνειο χωριστά, αυτό είναι τεράστιο πεδίο. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγουμε όσο γίνεται, για να μην πω πλήρως, περιοριστικές διατάξεις και υπερβολικά ε, ε, υπερβολικές ή Σας παραθέτω κάτι από ένα άρθρο του κανονισμού θα πρέπει να είναι τμήμα μιας δράσης με διαφορετικό επιλέξιμο ε, έξοδο, η δαπάνη Δηλαδή κάποιος ζητάει 10% επιδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά χρειάζεται και επιπλέον χρηματοδότηση εκτός από το 10% της επιδότησης. Να πάρει ένα δάνειο. Αν θέλει να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα του Ταμείου Εγγυήσεων, όπως είναι η πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Και τέλος, άλλη σύσταση. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την αυτονομία των εθνικών αρχών που μπορούν και να σχεδιάσουν τα χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική τους με νομική ασφάλεια, βεβαίως σε, πλήρη νομιμότητα, σεβόμενη και το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, χωρίς όμως αυτό το γκορσέ, τον υπερβολικό και χωρίς αυτές τις δρακόντιες διατάξεις. Οι συστάσεις λοιπόν, η πρωτοσολιτολισμοί αυτοί, έγιναν de facto νόμοι θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να έχουμε τη δυνατότητα με κάποια ασφάλεια και με κάποιες προϋποθέσεις και σεβόμενοι τον κοινοτικό νόμο να σχεδιάζουμε και εμεί χρηματοδοτικά μέσα και να μην περιμένουμε να έρθει ο κάθε οικονομικός ελεγκτής, λογιστής και να μας πει ότι αυτό δεν είναι επιλέξιμο και να μας το απορρίπτει. Αυτά είχα να σα πω και να μοιραστώ μαζί σα. Muchas ευχαριστώ πολύ. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω και κάποιους επισκέπτες που έχουμε ανάμεσά μας, εκλεκτούς επισκέπτες και αναφέρομαι uh, taking place in, the Parliament today and tomorrow. And... Επιτροπής των Σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση Χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ. Είμαι ο αντιπρόεδρος αυτής της Επιτροπής, όλα αυτά σας καλωσορίζω. Βλέπουμε ότι βυθιζόμεθα όλο και περισσότερο στον τόσο γοητευτικό κόσμο των χρηματοδοτικών μέσων και των άλλων τρόπων χρηματοδότησης. Η ομιλήτρια που θα πάρει τώρα τον λόγο είναι η κυρία Σουζάνα χάργητα η οποία θα μας δώσει μια συγκριτική παρουσίαση των χρηματοδοτικών μέσων από τη μία και των επιχορηγήσεων από την άλλη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την συζήτηση. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις στην απόψει τις οποίες έχει για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Για αυτούς που δεν μας γνωρίζουν καλά, είμαστε ένα διεθνές πιστοτικό όργανο, το οποίο έχει σαν στόχο τον ιδιωτικό τομέα, το 75% του χαρτοφυλακίου μας έχει σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε δραστήριοι στην κεντρική και ε, νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάποιοι από τις χώρες αυτές ε, έγιναν μέλη το 2004 και για περιορισμένο χρονικό διάστημα δραστηριοποιούμεθα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Έχουμε μια τιμολόγηση βασισμένη στις ε, τιμές της αγοράς ε, και επίσης ε, ελέγχουμε το θέμα της προσθετικότητας στις χώρες αυτές της Ένωσης που είμαστε μέλη. Η προσθετικότητά μας λειτουργεί σε σχέση με την διαθεσιμότητα ε, των άλλων μέσων όπως των περιφερειακών ταμείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων οπότε η προσθετικότητά μας είναι πολύ χαμηλότερη ε, χρηματοδοτούμε πάντως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως επίσης και το πέρασμα σε οικονομίες με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε δύο-τρεις ε, τομείς εκτός αυτών που αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι. Καταρχάς, χρειαζόμαστε ακόμα τις επιχορηγήσεις. Είναι κάποια θέματα τα οποία τίθενται και αναρωτιέται κάποιος αν έχει περάσει, αν θέλετε, ε, η μόδα των, των ε, επιχορηγήσεων προς την πλευρά μόνο των χρηματοδοτικών μέσων ιδιαίτερα για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Ένας από τους προηγούμενους μάλιστα είπε άραγε τα χρηματοδοτικά μέσα ή επιχορηγήσεις είναι υποκατάστατα μεταρρυθμίσεων της αγοράς και πώς τα δύο αυτά μπορεί να συμβιαστούν. Αλλά πριν περάσω στις 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια διαφορετική άποψη για τη χρήση των επιχορηγήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες το πώς ας πούμε χρησιμοποιούμε τη χρηματοδότηση αυτή στην Νοτιοανατολική Μεσόδιο, στα Δυτικά Βαλκάνια, εκεί ελέγχουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο με την Ένωση και έχουμε, είμαστε πιο επιλεκτικοί στους τομείς αυτούς και πιο στοχευμένοι από ό,τι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφοροποιούμε από το είδος της δραστηριότητας που χρηματοδοτούμε. Θα πρέπει να είναι εμπορική δραστηριότητα, διεύρυνση δημοσίων υπηρεσιών. Βλέπουμε σε ποιους τομείς μπορούμε να είμαστε παρόντες, ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται από την παρέμβαση αυτή. Έχουμε επίσης και κάποιες βασικές αρχές που χρηματοδοτούν την, τις επιχορηγήσεις τις οποίες δίδουμε εμείς στο σύνολο των χωρών μας, από το Μαρόκο μέχρι την Πολωνία, την Ουκρανία και την Κεντρική Ασία. Πρώτον πρέπει εμείς να αποφύγουμε να πιέσουμε τον ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει να αποδείξω στους μετόχους μου και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι <clears throat> έχουν γίνει όλες οι μελέτες των συνεπειών στην αγορά. Θα πρέπει επίσης να διαμορφώσουμε έτσι την χρήση των επιχορηγήσεων έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε εξαρτήσεις και θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα προγράμματα να δίδουν μακροπρόθεσμη οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα με δυνατότητα επιβίωσης με την δική τους δύναμη, τις δικές τους δυνάμεις. Έχουμε τις εσωτερικές μας κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση των επιδοτήσεων και των ευνοϊκών χρηματοδοτήσεων και για τομείς όπως το blending, η ανάμιξη μέσων και τέτοια θέματα καλύπτουν αν θέλετε τις λεγόμενες εξωτερικές εκθέσεις τις ατέλειες της αγοράς, θέματα διαθεσιμότητας, τα οποία τίθενται συχνά και επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τις νέες επιχειρήσεις και τις επενδύσεις υψηλού δυναμικού. Χρησιμοποιούμε λοιπόν εμείς τις επιχορηγήσεις και τις ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις με μετριοπάθεια και να μεγιστοποιήσουμε τις, τον, Now, going back... Τη μόχλευση για τις 12 ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες ε, λειτουργούμε πιστεύουμε ότι οι αρχές με τις οποίες λειτουργούμε ισχύουν και για τις υπόλοιπες ε, χώρες. Οι παρεμβάσεις μας είναι παρεμβάσεις οι οποίες δημιουργούνται μέσω προγραμμάτων που παράγουν έσοδα δηλαδή και σε κεφαλαιοποίηση, αύξηση διαθεσίμων και ε, μετάβαση σε οικονομική δραστηριότητα μειωμένων εκπομπών. Όπως βλέπουμε στο πολιετές πλαίσιο αναφοράς, στα λειτουργικά προγράμματα, ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε εκεί ένα επίπεδο που να γίνεται μια εκ των προσέρων αξιολόγηση και για τις επιχορηγήσεις και ε, για τα οικονομικά μέσα. Πολλές φορές ε, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 150 σελίδες. Πολλές φορές έχω διαβάσει τέτοιες αξιολογήσεις χωρίς συγκεκριμένες αναφορές σε στρατηγική, σε στόχους, σε λειτουργικές ανάγκες και πολλές φορές ε, ε, η ανάγκη ε, χρηματοδότησης, το τι θα επιλέξουμε για χρηματοδότηση ελείπει. Αυτό το οποίο βλέπουμε ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη είναι το να περάσουμε προς τα χρηματοδοτικά μέσα σε αυτές τις περιοχές και σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία κτλ βλέπουμε ότι οι διαχειριστικές αρχές έχουν ήδη μια δυσκολία στα πλαίσια της διαχείρισης των διαθεσίμων χρηματοδοτήσεων. Τα διαφορετικά μέσα έχουν και διαφορετικά επίπεδα περιπλοκότητας και συνεπώς διαφορετικούς κανόνες εφαρμογής τι είναι καλό και τι είναι κακό σε σχέση με τις επιχορηγήσεις. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι επιχορηγήσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο υποστηρίζοντας τις επενδύσεις όπου υπάρχει έλλειψη άλλου τύπου μορφών κάλυψης των οικονομικών αναγκών. Ιδιαίτερα δηλαδή σε τομείς όπου δεν παράγεται εισόδημα, δεν υπάρχει κέρδος από την επένδυση αυτή παρά μόνον έμεσα. Οι επιχορηγήσεις δίδουν πρόσβαση σε προγράμματα τα οποία από μόνα τους δεν μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτική ή δημόσια χρηματοδότηση. Εκεί βλέπουμε και κάποιες καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης και σε τομείς όπως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μπορούν επίσης να καλύψουν κάποιες συγκεκριμένες τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και να διευκολύνουν την έλευση επενδυτικών μέσων ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα ε, και όχι σε 5 ή 10 χρόνια. Και εδώ επανέρχομαι στο θέμα του περάσματος ε, στην οικονομία χαμηλών ποσοτήτων και χρήσεων άνθρακα. Ταυτόχρονα εμείς προσπαθούμε να σχεδιάσουμε ε, κάποια προγράμματα επιχορηγήσεων σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν και σε σχέση και με τις διαθέσιμες άλλες πηγές όπως τα χρηματοδοτικά μέσα ε, από διεθνείς και εθνικές επενδυτικές τράπεζες. Δεν είναι εύκολο όλα αυτά να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν. Όπως είπα, οι μεταφορές ωφελούνται από την χρήση των επιχορηγήσεων. Έχουμε δει μια σημαντική αν θέλετε, επιτάχυνση των διασυνδέσεων στον τομέα των μεταφορών, επίσης και περιφερειακών οδών και σιδηροδρόμων, αλλά όπως και θα πω πολλές φορές στη συνέχεια, αυτά είναι κάτι το οποίο μπορεί να προωθηθεί συνδυασμένα σαν παράδειγμα σωστή σχεδίαση των αναγκών στον τομέα των οδικών μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών, των εμπορικών σιδηροδρομικών μεταφορών και άλλων προγραμμάτων. Επίσης, ε, τμήμα των σημαντικών αυτών επενδύσεων θα πρέπει να είναι και η διαχείρισή τους μετά τη δημιουργία τους. Και επίσης ε, μπορεί κανείς ε, να χρησιμοποιήσει και μια έμεση ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε καλά παραδείγματα, σαν παράδειγμα στη Σλοβανία, Σλοβακία πόσο μπορεί να προωθηθεί η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην ενέργεια επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιχορηγήσεις για διαπεριφερειακές συνδέσεις ε, και διασφάλιση της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν δύο εβδομάδες πήραμε μέρος σε μια σημαντική ε, συζήτηση για τις προσθετικότητες που δημιουργούνται ε, στα πλαίσια των επιχορηγήσεων για την κοινή ενεργειακή πολιτική. Και οι επιχορηγήσεις εδώ είναι κάτι το οποίο θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από αυτούς οι οποίοι αναφέρονται κόστος, στην κατανομή του κόστους μεταφοράς ηλεκτρισμού. Κανένας δεν μπορεί να προσφέρει καλύτερη χρηματοδότηση από το διαθέσιμες στον τομέα αυτό επιχορηγήσεις. Τώρα στις τοπικές υποδομές έχει υπάρξει επιτάχυνση και στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά έχουμε όμως ε, μείνει πίσω σε σχέση με τον σχεδιασμό των πολιτικών που θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις στις πολιτικέ. Θα πρέπει να υπάρξει περιφερικοποίηση της διαχείρισης αυτών των ε, ε, δημοσίων, αν θέλετε, ή καθολικού τύπου υπηρεσιών μπορεί να υπάρξει ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα να παίξει ρόλο και στα πλαίσια της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ε, και επίσης να επιταχυνθεί η χρήση των επιχορηγήσεων για τις επενδύσεις. Τώρα στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, οι δύο τομείς τους οποίους έχουμε μείνει και έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η καινοτομία ε, η συγχρηματοδότηση για τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις και ο συνδυασμός με τα χρηματοδοτικά, τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα. Στην πράσινη οικονομία, στη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μετριοπάθεια και με σωστό έλεγχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οδηγεί στην απόσβεση του κόστους μεσοπρόθεσμα και είδαμε οι αγορές αυτές να εξελίσσονται προς τον τομέα αυτό σε χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία. Έχει υπάρξει μια συμμετοχή των επιχορηγήσεων γύρω στο 10 ε, με 12% και έχει επηρεάσει θετικά τη λειτουργία τους. Τώρα, ε, τι άλλο να πω για τα χρηματοδοτικά μέσα. Είναι πιο ε, περίπλοκα από τις επιχορηγήσεις και δεν θα πρέπει να είναι. Η δυσκολία η οποία υπάρχει είναι η διαχείριση των, ε, των μέσων αυτών και όχι τόσο η δημιουργία τους. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών μέσων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί και όχι και με καλύτερο τρόπο από ότι ας πούμε δικαιολογείται η δημιουργία και η χρήση των επιχορηγήσεων μέχρι τώρα. Θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα, θα πρέπει να δίδουν εγγυήσεις για περαιτέρω χρηματοδότηση και θα πρέπει να δίνουν ακριβώς την δυνατότητα κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη τα μέσα αυτά βρίσκονται σε εφηβική ηλικία. Όχι μόνο γιατί απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, αλλά και ικανές εφαρμοστικές δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι χώρες οι οποίες είναι πιο έμπειρες στη χρήση αυτών των μέσων έχουν ισχυρές περιφερειακές τράπεζες, ενδιαμέσους κτλ. Και δεν είναι τυχαίο ότι το εθνικό επίπεδο χρηματοδοτικών μέσων φαίνεται να λειτουργεί και να σχεδιάζεται καλύτερα σε υποπεριφερειακό επίπεδο. Να αναφερθώ επίσης δύο σε δύο τομείς, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολία στη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Το ένα είναι οι εγγύησει παράλληλα με τις επιχορηγήσεις. Κάποιοι από τους προηγούμενους ομιλητές είπαν ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παράλληλα προγράμματα για την, μικρο, για την χρηματοδότηση των μικρών μεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων. Ένα τομέα τον οποίο θα θέλαμε εμείς να προωθήσουμε είναι το λεγόμενο streamlining του ευρωπαϊκού επίπεδου λειτουργίας των χρηματοδοτικών μέσων και του εθνικού, γιατί υπάρχει ένας κάποιος κανιβαλισμός στην αγορά κεφαλαίου γύρω από τα θέματα αυτά. Υπάρχουν κάποια προγράμματα επιχορηγήσεων που λειτουργούν παράλληλα με τα χρηματοδοτικά μέσα και αυτό δημιουργεί δύσκολες δυνατότητες επιλογής για το ποια είναι η προτιμητέα λύση. Για τις μικρομεσαίες λοιπόν είναι δύσκολο και είναι δύσκολο και για τις κυβερνήσεις να υπολογίσουν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών. Ένας άλλος τομέας στον οποίο έχουμε βρει ε, μια ε, πολύ μεγάλη δημιουργία ε, <clears throat> τέτοιου είδους επενδυτικών μέσων είναι η διασφάλιση ρευστότητας. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ε, τις δυναμικές της αγοράς κάθε φορά. και υπάρχει ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση σε τομείς με υψηλή επιτάχυνση και δύσκολη έβρεση πόρων μέχρι τώρα. Θα πρέπει να επιλέγονται σωστοί διαχειριστές όμως με μεγάλη εμπειρία για τη διαχείριση αυτού του είδους των ενεργειών είναι σαν στόχος κάτι τοποθετικό, αλλά η επιλογή του διαχειριστή είναι κάτι το πολύ πιο σημαντικό αν θέλουν να αναπτύξουν τις αγορές αυτές ε, κεφαλαίων και όχι μόνο να διασφαλίσουν μια εφάπαξ ενίσχυση κεφαλαιοχική. Ε, Υπάρχει επίσης ε, και συγκεκριμένη αναφορά στις ε, διαθέσιμες επενδυτικές δυνατότητες στις αγορές όπως επίσης και τις μικρομεσές οι οποίες έχουν χαμηλά επίπεδα ιδίων κεφαλαίων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οι ε, σύμβουλοι να είναι σε θέση να επιλέξουν σωστά. Θα πρέπει να μπορούν να κάνουν επενδύσεις σε εταιρείες στις οποίες ε, υπάρχει έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, αλλά αυτό μόνο του σαν κριτήριο δεν αρκεί. Από την εμπειρία μου αναφέρθηκα ήδη πως μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε και με τα θέματα των αξιολογήσεων εξάντε που εν πολλής ήταν άχρηστες οι αξιολογήσεις αυτές, τουλάχιστον αυτές που διαβάσαμε. Δεν περιελάμβαναν συστάσεις για τον τρόπο κατά περίπτωση σχεδιασμού των χρηματοδοτικών μέσων δεν έχουν κρίνει και να βοηθήσουν να υπάρξει η διάκριση ανάμεσα στα χρηματοδοτικά μέσα και τις επιχορηγήσεις. Να πω ότι οι επιχορηγήσεις οι επενδύσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και με μεταρρυθμίσεις στον τομέα των πολιτικών. Να μην μιλήσω εδώ για αιρεσιμότητα, αλλά η βασική ιδέα είναι ότι υπάρχει πολλές φορές ε, μια σταδιακή διαδικασία χρήσης ε, και των διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. <clears throat> Και θα πρέπει επίσης ε, να μην λειτουργούμε μόνο για να προστατεύουμε αν θέλετε τις επενδύσεις αλλά να προσκαλούμε τα χρηματοδοτικά μέσα και τις διαθεσιμότητες της εμπορικές να επενδύουν σε στοχευμένους τομείς δύο επιπλέον θέματα. Πρώτον, θα πρέπει να σχεδιάζεται προγράμματα επιχορηγήσεων με τεχνική βοήθεια, με τεχνική αρρωγή. Όταν μιλάμε με τις εθνικές επενδυτικές τράπεζες ή με τα κατά μία, πολλές φορές λέγουν ότι δεν έχουν τη διάθεσή τους την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται. Τώρα όμως είναι βασικό αυτό να γίνει όχι μόνο για τον σχεδιασμό αλλά και για τη βελτίωση της ικανότητας του τελικού ε, εποφελούμενου από τα ποσά αυτά να τα διαχειριστεί. Αναφέρομαι και σε εταιρείε εδώ διαχείρισης στερεών αποβλήτων και σε μικρομεσαίες που σχεδιάζουν προγράμματα και σε ενίσχυση των θέσεων των ενδιαμέσων ε, χρηματοδοτών και για τα προγράμματα ε, τα υπόλοιπα στα οποία η έλλειψη τεχνικών γνώσεων δημιουργεί θέματα. Πολλές ιδέες έχουν κατατεθεί στον τομέα αυτό, πάντως ε, έχω αναφερθεί σε κάποιες από αυτές τις ιδέες που θα θέλαμε να υπάρξουν αλλαγές. Εμείς συζητάμε με τις διαχειριστικές αρχές στις 12 χώρες αυτές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης όπου είμαστε παρόντες τι γίνεται Είχαμε πρόσφατα μία συνάντηση με συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα εξωτερικών επενδύσεων και συζητήσαμε το θέμα των εγγυήσεων και εδώ έχουν κατατεθεί ορισμένε νέες ιδέες σε σχέση με τον έλεγχο της χρήσης των δημόσιων πιστώσεων για την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Πάντως πιστεύουμε ότι η εμπειρία την οποία θα έχουμε σωρεύσει και με το πρόγραμμα εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης αλλά και εσωτερικά. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να ακούσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα ήθελα Καταρχάς, ε, να δώσω το λόγο στην κυρία Συγγετρία, παρακαλώ. Ε, κυρία Καρδιεθάμπαλ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση εγώ, την οποία έγραφα ε, ακούγοντας τους ομιλητές. Αν και η κυρία Χαρκιτάη εν μέρει απάντησε. Λοιπόν, ακούγοντας αυτό που μας λέτε για τα προϊόντα ή τα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιείτε, Λέτε ότι ορισμένα δεν λειτουργήσαν πολύ καλά, ήταν πολύ περίπλοκα και η ΚΑΕΦΒ μας μίλησε για το πολιτισμό, τις δημιουργικές βιομηχανίες. Σύμφωνα με την πείρα σας, ποια είναι τα χρηματοδοτικά μέσα και προϊόντα που θα πρέπει να διατηρήσουμε, να τα κρατήσουμε και ποια να καταργήσουμε ακριβώς επειδή δεν αποδίδουν ή να τα ξανασκεφτούμε στο μέλλον, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια στους τομείς που αυτή τη στιγμή συζητούμε και τις πολιτικές στις οποίες έχουμε παρεμβάσεις, πού θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή η συμμετοχή των χρηματοδοτικών μέσων, γιατί αυτή η έλλειψη χρηματοδότησης και επενδύσεων παραμένει τεράστια και οξύτατη και δεν μπορούμε να βρούμε ε, χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες δηλαδή. Πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, Έιντερ. Σε ποιον απευθύνονται οι ερωτήσεις. Α, σε όλους. Δεν υπάρχει θέμα. Ε, για λόγους σαφήνειας θα ήθελα να κάνετε μία ερώτηση ε, ο καθένας ε, και να λέτε σε ποιον απευθύνεται για να απαντά. Ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος στην ερώτηση της εισηγητρίας. Some, somebody cast the first stone, please. I will give it a shot. Θα προσπαθήσω εγώ. Καταρχάς, ένα από τα πράγματα που προσπάθησα να πω είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά μέσα για κάτι πολύ συγκεκριμένο, για παράδειγμα, για τους δημιουργικούς τομείς. Μπορεί να θέλει να παρέχει κανεί ε, χρηματοδοτικά μέσα σε επιχειρήσεις, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μερικές από αυτέ ε, δραστηριοποιούνται στο δημιουργικό τομέα, άλλες όχι. Μπορεί λοιπόν ε, να θεωρήσει κανείς ότι είναι καλή ιδέα αυτή, αλλά εγώ δεν θα δημιουργούσα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για αυτές. Επίσης, Είπαμε ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα εργαλεία και η ενεργειακή απόδοση είναι μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν τόσο πολλά κτίρια, τόσο πολλά θέματα, τόσα προβλήματα που πρέπει να λυθούν μεταξύ ε, ενοικιαστών και εκμισθωτών ε, και όσον αφορά τα αστικά ταμεία και ε, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αποτελεσματικά. Κάποιοι λένε ωραία, έχουμε χρηματοδοτικά μέσα για τις πόλεις, σας κάνουμε κάτι τώρα και για, το, και για τις ε, αγροτικές περιοχές. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Μπορεί να φανταστώ κάποιου τομεί, αλλά να δημιουργήσουμε χρηματοδοτικά μέσα για οπουδήποτε και επειδή κάτι λειτουργεί για τα κτίρια, να θεωρήσουμε ότι θα λειτουργήσει και στι αγροτικέ περιοχέ, αυτό νομίζω ότι είναι αφελέ. Φαντάζομαι ότι μπορεί κανείς ε, να δημιουργήσει επιχειρήσεις ε, εκμεταλλεύσεις ε, στη γεωργία που να μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην νομίζουμε ότι ταιριάζει παντού κάτι τέτοιο. Και η βασική μου σύσταση δεν είναι να επικεντρωθούμε υπερβολικά. Και επίσης βλέπουμε έναν τομέα που μπορεί να αναπτύσσεται συνεχώς Μπορεί να υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη κάποια στιγμή όμως να ε, τα πάει τόσο καλά ο τομέας ε, ώστε να μην ε, έχει πια ανάγκη τις τράπεζες και τα δάνεια. Τα πράγματα αλλάζουν. Σε δύο χρόνια μπορεί κάποιος τομέας να αποφετήσει εδώ σαν να μην χρειάζεται πια χρηματοδοτικά μέσα. Αυτά ήθελα να πω και να δώσω το λόγο σε οποιονδήποτε μπορεί να προσθέσει κάτι ή να βελτιώσει αυτά που είπα. Η κυρία Χάρκιτάη, παρακαλώ. Κάποιες ιδέες, αλλά ακολουθώντας λίγο πολύ τις ίδιες γραμμές. Τέσσερα πράγματα. Καταρχάς είδαμε πάλι την χρήση του πιο επικίνδυνου χρηματοδοτικού μέσου, της ε, εγγύησης για την ε, πρώτη απώλεια. Και οι τράπεζες ε, μπορεί να έχουν όρεξη για κίνδυνο. Ένα τέτοιο μέσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. αλλά ε, μας λείπει η χρηματοδότηση ε, χρεών υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη όρεξη στις τράπεζες να μπουν στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου που χρειάζονται αρχική υποστήριξη. Επίσης, ε, είπα ότι χρειάζονται ακόμα κεφαλαϊκές επενδύσεις ε, για επιταχυντές ε, που υποστηρίζουν την καινοτομία δηλαδή. Ο τρίτος τομέας αναφέρθηκε και από τον Χόρχε. επιχειρηματολογήσαμε κατά ενό χρηματοδοτικού μέσου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, που θα είχε όμως να κάνει με την ε, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η ηλιακή η αιωλική ενέργεια μπορεί να μην χρειάζονται περαιτέρω ε, επενδύσεις υψηλού κινδύνου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν εγγυήσεις και σε πλατφόρμες εθνικές και τοπικές για επενδύσεις, ώστε να χρηματοδοτηθεί να χρηματοδοτηθούν μαζικά ε, προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Και βέβαια το ορφανό παιδί όλων μας ε, είναι οι αγροτικές επιχειρήσεις, ε, το agrobusiness. Ο καθένας σκέφτεται τον αγρότη που πεινάει, αλλά και πάλι έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Νομίζω όμως ότι η Ευρώπη έχει μείνει στο, πίσω στο θέμα αυτό και ιδιαίτερα η Ανατολική Ευρώπη. Να έχουμε δηλαδή βιώσιμα χρηματοδοτικά μέσα που να μπορέσουμε να ε, σπρώξουν την γεωργία προς τον τομέα της επιχειρηματικότητας. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ αρκετά με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Για να είμαι ειλικρινής, αν δούμε τα μέσα που προσπαθούμε τώρα να στήσουμε τη συγκεκριμένη περίοδο, ένα από αυτά και ίσως το μοναδικό όπου θα έμπαινε το κράτος για όλη τη χώρα είναι αυτό για την ενεργειακή απόδοση και στις κατοικίες, δηλαδή ε, στους ιδιώτες, αλλά και στις επιχειρήσεις. Εκεί υπάρχουν και ανάγκες και ανάγκη χρηματοδότησης. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ιδιωτική κατοικία το θέμα είναι περίπλοκο. Σε κάποιες χώρες όπως η Ισπανία όπου ο περισσότερος κόσμος ε, ζει σε κάποιες πολυκατοικίες ή ε, συνειδιοκτησίες. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ άκαμπτη. Πολλές φορές χρειάζεται ομοφωνία όλων των ενίκων και είναι αρκετά περίπλοκο ε, να γίνει αυτό. Για τις επιχειρήσεις είναι πιο εύκολο. Είχαμε μια καλή εμπειρία με το Μέσω που άρχισε το 2007 με 2013 έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και σχεδόν ε, έχουμε καταλήξει εμείς να χρηματοδοτούμε ε, έργα του ιδιωτικού τομέα. Άρχισε αυτή η επιχείρηση για τα δημόσια κτίρια και κατέληξε να χρηματοδοτούμε <laughs> ιδιώτες. Και ακόμα δεν έχουν ε, ε, πραγματική ουσιαστική παρουσία οι εταιρείε αυτές ε, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα. Συμφωνώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να σχεδιάσουμε χρηματοδοτικά μέσα για κάθε ειδικό ή συγκεκριμένο τομέα. Αλλά για τύπο χρηματοδότησης, αναφέρθηκε εδώ το κεφάλαιο κινδύνου. Εκεί πραγματικά υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ανάγκη της χρηματοδότησης αυτών των ε, επιχειρήσεων. Στην Ισπανία Εκεί που χρειάζεται κάλυψη περισσότερο κεφαλαίου κινδύνου είναι εκεί που δεν χρηματοδοτούμαστε από τα ε, διορθωτικά ταμεία. ή τα διαρθρωτικά ταμεία με την παραδοσιακή ε, μορφή δεν υπαρκούν. Και θα μπορούσε αυτό να είναι και τραυματική εμπειρία για τον προπολογισμό μας. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ανάγκη χρηματοδότηση, αλλά και πού και τι χρηματοδότηση Γι' αυτό χρειάζεται ενδεχομένω μεγαλύτερη ευελιξία σε εθνικό επίπεδο. Για να μπορεί να καλύπτεται όλη η επικράτη. Αλλιώ ίσως έχουμε πρόβλημα. Από άλλα μέσα που δεν υπάρχει συγχρηματοδότηση και συνυπευθυνότητα βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια ανισορροπία αρκετά μεγάλη μεταξύ περιφερειών. Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε πόρους, αλλά πολλές φορές δεν είναι αρκετά ποιοτικά τα έργα για να είναι επιλέξιμα. Ας πούμε, για τη χρηματοδότηση καινοτομία ή ε, το, ένα κεφάλαιο έναρξης ε, μιας επιχείρησης. Το αρχικό κεφάλαιο. Τι συμβαίνει εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σχεδιάσουμε την κατάλληλη μέθοδο διαχείρισης κάθε χρηματοδοτικού μέσου. Στην προηγούμενη περίοδο εμείς δρομολογήσαμε ένα χρηματοδοτικό μέσο για καινοτόμες επιχειρήσεις. Για όλους τους τομείς διακλαδική, αλλά μέσω ενδιάμεσων οργανισμών που δεν λειτουργήσε το σύστημα. Γιατί με τα προπετούμενα που θέσαμε ε, για την πιστοποίηση, για τον έλεγχο, ο κλάδος ε, της ε, χρηματοδοτικός δηλαδή, οι ενδιάμεση δεν ενδιαφέρθηκαν. Τώρα μπορείς να επιλέξεις ως ενδιάμεσο μια αναπτυξιακή τράπεζα που ε, θα έχει ως σκοπό να ενισχύει τις κοινοτόμες επιχειρήσεις. Αυτό έχει νόημα γιατί είναι και ο λόγος ύπαρξης της συγκεκριμένης τράπεζας ή του συγκεκριμένου ιδρύματος. Πολλές φορές λοιπόν αυτό που φταίει δεν είναι η θεωρία το πώς θα είναι το μέσο αλλά πώς έχει σχεδιαστεί πρακτικά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. να δώσω το λόγο στον κύριο Τεκόφσκι στα δεξιά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευγνώμων για τη σημερινή συζήτηση. Ε, χαμογέλασα ακούγοντας κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν. Η Επιτροπή μας συχνά επικρίνει κάποια μέτρα που λαμβάνονται με τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις αυτές. Είπατε ότι τα χρηματοδοτικά μέσα στηρίζουν νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν μπορούν να λάβουν μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική υποστήριξη. Και είπατε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται και να διατηρούν προγράμματα μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι αυτό είναι πράγματι πρόβλημα. Επί 13 χρόνια ασχολούμαι με νεοφυείς επιχειρήσεις και κοιτώντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις που στηρίζονται με μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπω ότι δεν έχουν λογική, δεν έχουν επιχειρηματικό σχέδιο, δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Ε, δεν ε, ζουν πάνω από τρία χρόνια αυτές οι επιχειρήσεις. λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τα τυπικά προσόντα, τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιχείρησης, όχι όμως τον αντίκτυπο. Ανταποκρίνονται οι αγορές. Για παράδειγμα, μπορεί μια νεοφύση επιχείρηση να ε, έχει μια εξαιρετική ιδέα. Εάν όμως δεν λάβει δίπλωμα ευρυστεχνίας για αυτήν την ιδέα, μπορεί κάποιος άλλος να την αντιγράψει. Και έτσι να πηγαίνει χαμένη όλη η υποστήριξη που τους δώσαμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα μπορεί να είναι η επιλογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται. Για παράδειγμα, στην Τσεχία χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό όμως δεν ε, λύνει το πρόβλημα της Πολωνίας που είναι αντίστοιχο. Για παράδειγμα, μπορεί να, να χτίζουμε έναν δρόμο στην Τσεχία μέχρι τα σύνορα, να μην υπάρχει όμως συνέχεια από την πολωνική πλευρά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει με έργα στην Ισπανία και αλλού. Κατόπιν υπάρχει το γενικό πρόβλημα ότι κάποιες τράπεζες έχουν τεράστιες χρηματοδοτικές δυνατότητες, δεν επενδύουν όμως και κυρίως δεν επενδύουν σε προγράμματα που ε, να έχουν κάποιον κίνδυνο ή τουλάχιστον όχι τόσο όσο στο παρελθόν. Για παράδειγμα, στον τομέα της στέγασης δεν είναι ανταγωνιστικές με κάποια είδη χρηματοδότησης που παρέχονται. Για παράδειγμα, η οικογένειά μου είχε ένα μεγάλο σπίτι από τη δεκαετία του 30. Ε, πρόκειτο για κοινωνικές κατοικίες, ήταν λοιπόν ένα μεγάλο κτίριο γεμάτο μικρά διαμερίσματα. ο ιδιοκτήτης ε, μπόρεσε να χρηματοδοτήσει άλλα προγράμματα με αυτά τα μικρά διαμερίσματα. Τώρα ε, μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης με τα ταμεία συνοχής, αλλά είναι πολύ δύσκολο στον τομέα της στέγασης να δοθεί η ευκαιρία για παρόμοια έργα. Ας σκεφτούμε λοιπόν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην δημιουργείται ανταγωνισμός που να υπονομεύει οι παραδοσιακές πρακτικές ε, στις διάφορες χώρες. Αυτή είναι η θέση μου που ήθελα να σας παρουσιάσω. Θα εκτιμούσα αν μπορούσατε να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα αυτά. Επίσης αναφέρθηκαν διάφορες χώρες, ε, αλλά εγώ γελάω που τα ακούω, διότι σε πολλές χώρες υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν εάν δεν υπάρχει σωστή επιβολή του νόμου, εάν χαθούν τα χρήματα, εάν τριπλασιαστούν οι τιμές. Ε, είναι πολύ δύσκολο να παράσχει κανείς βοήθεια. και οι δυνατότητες μόχλευσης κάποιων τέτοιων προγραμμάτων ήταν ουσιαστικά μηδενική. Η αμεληταία σε σχέση με προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν με εμπορικά κεφάλαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε διάφορα προβλήματα. Θα ήθελε κανείς να σχολιάσει. δεν ε, βλέπω πολύ προθυμία. Πολύ σύντομα να συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση και να προσθέσω ότι εάν χτιστεί δρόμος σε κάποιο κράτος μέλος χωρίς ε, να λαμβάνονται υπόψη από την αρχή οι ευρωπαϊκές συνέργειες, αυτό δεν επιφέρει απαραίτητα ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. το να ε, παραταθεί ο δρόμος από την άλλη μεριά των συνόρων εάν δεν είχε ληφθεί από την αρχή υπόψη η ευρωπαϊκή διάσταση που θα μπορούσε να είχε. Παρακαλώ. Ήταν ε, μακρύς ο κατάλογος ε, των θεμάτων ε, και όπως και οι επιχορηγήσεις, έτσι και τα χρηματοδοτικά μέσα, ε, λειτουργούν ανάλογα με το πόσο καλά λειτουργούν ε, οι φορείς εφαρμογής. Μπορεί να έχουμε έναν δρόμο που να οικοδομηθεί, αλλά στα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα και αυτό μπορεί να αποτελεί κίνητρο. Εάν δεν μπορέσει να ανακτήσει κανείς τους πόρους που επένδυσε, ε, τότε αυτό είναι πρόβλημα. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να γίνει αυτό είναι αν έχουμε έναν δημόσιο φορέα που να ε, αποπληρώνει το δάνειο. Δηλαδή έχουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο και κάποιος δημόσιος φορέας ε, αποπληρώνει το δάνειο και μπορεί έτσι να κάνει διάφορα έργα. Ε, η κακή εφαρμογή λοιπόν δημιουργεί προβλήματα και αυτό είναι ένας λόγος που δεν βλέπουμε χρηματοδοτικά μέσα σε όλες τις χώρες και δεν βλέπουμε να διαδίδονται περισσότερο διότι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες σε κάποιες χώρες. Ε, άλλες χώρες είναι πιο προηγμένες, ε, έχουν και καλή διαδικασία επιλογής. Εγώ λοιπόν δεν θα κατηγορούσα τα χρηματοδοτικά μέσα, θα κατηγορούσα αυτούς που εγκρίνουν τα προγράμματα. Αυτά. Ευχαριστώ να μιλήσω και εγώ για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το τι είδους επιχειρήσεις προσπαθούμε να στηρίξουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιους στηρίζουμε στην KFW. Στηρίζουμε με, διάφορα, με διαφόρων ειδών ε, χρηματοδοτικά μέσα, διαφόρων ειδών ε, νεοφυείς επιχειρήσεις. Μπορεί να έχουμε ε, ιδιαίτερα καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις όπου δίνουμε επιχορήγηση στις πολύ καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουμε ε, προγράμματα επενδύσεων υψηλού κινδύνου. Μπορεί να δομήσει λοιπόν κανείς ανάλογα τα χρηματοδοτικά μέσα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το πολιτικό πλαίσιο είναι πολύ βασικό και θα ήθελα να πω ότι έχουμε προγράμματα και στη Βόρεια Αφρική και σε χώρες όπου είναι πολύ χειρότερο το πολιτικό πλαίσιο από αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι τα διάφορα είδη χρηματοδοτικών μέσων ε, πρέπει να προσαρμοστούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Είτε θέλεις να σχολιάσεις? Όχι. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα να καλέσω την εισηγήτρια να συνοψίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να συνοψίσω, δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να βγάλω τα συμπεράσματα. Κάποιες σκέψεις, αν θέλετε, να μοιραστώ μαζί σας και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναλύουμε το θέμα και στο μέλλον και κάποιες από τις απαντήσεις που λάβαμε, τις μη απαντήσεις μάλλον, τι εννοώ. Όταν αναθέσαμε τη μελέτη στη ΣΕΠΣ ε, για να ε, κάνουμε τη συγκεκριμένη σημερινή ακρόαση για τα χρηματοδοτικά μέσα, ο σκοπός μας ήταν να δούμε αν μπορούμε κάπως να συστηματικοποιήσουμε τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, από τη μια τις επιχορηγήσεις και από την άλλη τα δάνεια ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Και αν μπορέσουμε να ορίσουμε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται κάθε φορά για να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο ή όχι, καλώς. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν συστηματικοποιείται αυτό, από ό,τι ακούμε. Εξαρτάται πάρα πολύ από τη χώρα, από τον κλάδο, ακόμα και από τους ε, ενδιάμεσους που χρησιμοποιεί κανείς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή αν μπορούν να συνδυαστούν με διαρθρωτικά ταμεία. Δηλαδή αυτή η συστηματικοποίηση, ο πίνακας που είχα στο μυαλό μου μάλλον δεν γίνεται. πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στην ιδέα να είναι πιο ευρύς ο ορισμός της χρήσης των χρηματοπιστωτικών μέσων. Το κατανοώ απολύτως. Ε, δεν θα πρέπει να είναι τόσο περιορισμένο το πεδίο εφαρμογή ή συγκεντρωμένο. Αλλά εμείς πολλές φορές οι πολιτικοί θέλουμε να καθοδηγήσουμε προς ε, κάποια πολιτική ε, τη δράση μας. Και δεν ξέρουμε πότε είμαστε ιδιαίτερα περιοριστικοί, πότε έχουμε περισσότερο ε, χώρο ή περιθώριο λιγμών. Και εδώ αναφέρομαι στις στους κλάδους της δημιουργίας και της πολιτιστικής παραγωγής για να μπορούν να χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όταν το μέσο είναι τόσο περιορισμένο και τόσο περιοριστικό, χάνουμε το στόχο μας. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια χρυσή τομή μια ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική κατεύθυνση που θέλουμε εμείς να δώσουμε για το πώς θα τα δημόσια χρήματα και το ποιο θα ενισχύσουμε ε, αυτή είναι λοιπόν η αρετή που είναι το ζητούμενο. Ε, τώρα για τα προαπαιτούμενα. Είναι γεγονό ότι τα περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα χρηματοδοτούν έργα τα οποία υποτίθεται ότι θα έχουν οικονομική απόδοση για την αποπληρωμή. Και από μόνο του αυτό είναι θετικό. Και δεν θα έπρεπε εμεί να έχουμε τόσα προαπαιτούμενα και τόσε απαιτήσει γενικότερα ή τόσα διοικητικά εμπόδια γιατί τελικά θα αποπληρωθεί αυτό το δάνειο, αλλά παραμένουν οι πόροι δημόσιοι. Οπότε φυσικά άλλο είναι η επιχορήγηση και άλλο το χρηματοδοτικό μέσο, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπως είναι οι εγγύησεις όπου τα δημόσια χρήματα μπορεί να χαθούν εκεί. Γιατί χρηματοδοτείς ένα έργο το οποίο πήγε στραβά ή για κάποιο λόγο δεν αποπληρώνεται. Άρα θα είναι βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δηλαδή δεν είμαστε στην επιχορήγηση και στις αντίστοιχε απαιτήσει, αλλά επειδή είναι δημόσια τα χρήματα και παραμένουν, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να τηρούνται. Αυτό έχει μεγάλη σχέση με αυτό που είπαμε προηγουμένως γιατί είναι εκ των προτέρων αξιολόγηση. Θυμάμαι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όταν προετοιμάζαμε τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, τις παρούς δηλαδή, ε, δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στην εκ των προτέρων αξιολόγηση. Αλλά τελικά τι είδαμε, ότι την κάναμε τόσο σημαντική ώστε έγινε αναποτελεσματική ως μέσο. Και είναι μάλλον ε, ε, γραφειοκρατικό και διοικητικό εμπόδιο παρά πραγματικό έγγραφο ενημέρωσης που θα μπορεί να μας επιτρέπει να επιλέξουμε το χρηματοδοτικό μέσο που ενδείκνεται για το συγκεκριμένο έργο. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πιο αρμόδια για αυτά τα θέματα. Μαζί μας βέβαια. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο Χόρχε Νούνιεθ Φερέρ, να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα κοινό έντυπο, ένα format, όλοι να δίνουν τις ίδιες πληροφορίες για να μπορούν αυτά τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα. Κάτι άλλο που ακούσαμε επανειλημμένος και είναι εύστοχο και εδώ επέμειναν πολλοί ομιλητέ, είναι η ανάγκη να διευκολυνθεί ή ο συνδυασμός αυτών των δύο επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων. Γιατί στα χαρτιά μπορεί αυτό να είναι δυνατόν, αλλά στην πράξη είναι τόσο περίπλοκη ο συνδυασμό αυτων των δυο επιχορηγησεων και χρηματοδοτικων μεσων γιατι στα χαρτια μπορει αυτο να ειναι δυνατον αλλα στην πραξη ειναι τοσο περιπλοκη η κατασταση οι απαιτήσει και τα κριτήρια και τόσο αντιφατικά που κάποια στιγμή να βαγεί αυτή η προσπάθεια. Αυτό το θέμα της απλούστευσης το έχουμε δει και εμείς στο δημοσιονομικό κανονισμό. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε, δεν ξέρω αν το καταφέραμε. Θα δούμε τι θα βγει από τις διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό κανονισμό. Είναι γεγονός πάντως ότι ένας από τους στόχους ήταν η απλοποίηση ακριβώς. Γιατί έχουμε πλήθος κανόνων που δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυαστούν. Άλλο, να βελτιώσουμε λέτε τον ορισμό αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Ιδιαίτερα στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και των στόχων για να αποφύγουμε επικαλύψεις των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό το είδαμε και όταν ξεκίνησε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είχαμε κάποιες επικαλύψεις με άλλα ταμεία. Με το Horizon 2020 ή με την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη ή το COSME. Κάποια στιγμή έχουμε ένα συνοθήλευμα ε, μέσων που συνδέονται μεταξύ τους, επικαλύπτονται και δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Ευελιξία. Αυτό είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας ανεξαρτήτως θέματος, αλλά δεν καταλήγουμε στην ευελιξία να την ορίζουμε με το σωστό τρόπο. Εδώ λέτε ευελιξία για να μπορούμε να εφαρμόζουμε και να προσαρμόζουμε στην πράξη ε, τα χρηματοδοτικά μέσα, σεβόμενοι την εκάστοτε πραγματικότητα της κάθε χώρας, μέλους ή περιφέρειας. Για να δούμε, θα την επιτύχουμε αυτή την ε, ευελιξία. Σημείωσα επίση και το θέμα αυτό της τεχνικής βοήθειας, πολύ σημαντικό. Ανέκαθεν αναφέραμε την ε, ανάγκη αυτή τεχνικής βοήθειας για να δημιουργηθεί η ικανότητα ε, απορρόφησης και εκτέλεση αυτών των πόρων και των χρηματοδοτικών μέσων. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος ξέρει την ύπαρξή τους, αλλά αγνοεί τη λειτουργία του ή το πώ θα μπορέσει να λάβει την τεχνική βοήθεια για να βελτιώσει την ικανότητα απορρόφησης. Εν πάση περιπτώσει και τελειώνω. Έλεγα στην αρχή ότι δεν απάντησαν στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Όχι επειδή δεν θέλησαν, αλλά επειδή δεν έχει μάλλον απάντηση αυτό. Υπό την έννοια ότι για την επόμενη θητεία θα πρέπει να αποφασίσουμε από τώρα ποιο θα είναι το ποσό που θα αφιερωθεί στα χρηματοδοτικά μέσα και ποιο θα είναι το ποσό που θα αφιερωθεί στις επιχορηγήσεις για κάποιες δημόσιες πολιτικές. Εκεί θα γίνει. Ο Καυγάς εκεί θα δοθεί η μάχη. Έχουν και τα δύο τους υποστηρικτές τους και τους πολέμιους το πεδίο διευρύνει τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να επιτύχουμε αυτόν τον τετραγωνισμό του κύκλου, αλλά αυτά είναι για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Πολύ μετριοπαθή είσαι. Ε, ότι ήταν, ήταν πολύ εξαντλητική η τοποθέτηση και τα συμπεράσματα. Λοιπόν, εξονο... Από πλευρά μου τώρα, να πω ότι έχει σημασία για την Επιτροπή μας να κατανοήσει όσο είναι εφικτό τουλάχιστον. Την ιδιαίτερα περίπλοκη φύση των χρηματοδοτικών μέσων και σήμερα χάρη στις εξαιρετικές σας παρουσιάσεις και την προετοιμασία σας, να σας συγχαρώ γι' αυτό. Μορφωθήκαμε Ακούσαμε στην αρχή τι είναι τα μέσα αυτά, πώς δημιουργούνται, αλλά ακούσαμε και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, πότε να τα χρησιμοποιούμε και σε ποιο τύπου περίπλοκες καταστάσεις να τα προτιμούμε. Ακούσαμε τις απόψεις μιας εθνικής επενδυτικής τράπεζας όπως από τη Γερμανία Ακούσαμε αρκετή κριτική από την οποία συγκρατώ το ότι, ότι πράγματι θα πρέπει εμείς να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο να ξεκαθαρίσουμε λίγο την απαράδεκτη κατάσταση των επικαλύψεων και των επικαλυπτόμενων κανονισμών. Καυκικές καταστάσεις όπως τις είπατε, αδικαιολόγητες εντελώς διακανονιστικές μορφές περιορισμών. Είναι αρκετά σκληρή η κριτική αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι τεκμηριωμένη. Ακούσαμε και τις δυσκολίες στη χρήση των μέσων, δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, τη χρήση των εγγυήσεων παράλληλα με τα προγράμματα επιχορηγήσεων και κάτι για το οποίο κάτι θα πρέπει να κάνουμε είναι η έλλειψη έμπειρων διαχειριστών των μέσων αυτών, των ταμείων αυτών, τους οποίους πράγματι χρειαζόμαστε και πρέπει να έχουμε σε μεγαλύτερους αριθμούς. Αυτά ήταν νομίζω μια χρήσιμη συνάντηση. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον καθένα σας και όλους μαζί για την εξαιρετική σας προετοιμασία. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνάντηση αρχίζει αύριο στις 9 το πρωί.